Καλημέρα συνάδελφοι, λέει ο κύριος Στάς. Α, τώρα είμαστε τέσσερις. Αντί για δύο οι ευρωβουλευτές. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τις εργασίες μας. Καλώς ορίσατε. Το πρώτο μας θέμα είναι η έγκριση της ημερήσης διάταξης. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Δεύτερον, ανακοινώσει του Προέδρου. Σήμερα για τελευταία φορά προεδρεύω γιατί ο σύνδεσμος ε, ακόμα έχει την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή αλλά έπρεπε να παρήσατε στην ε, Νάπολη για κάποια υπουργική συνάντηση. και θα αντικατασταθεί κάποια στιγμή εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε από τους φιλελευθέρους θα προέλθει ο νέος μας ε, πρόεδρος αρχέ. Ιουλίου. Μπορείτε να δείτε στο κοκομπού info τις ε, γλώσσες ε, στις οποίες θα εργαστούμε και επίσης μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και για να ακούγεται καλά η φωνή σας να μιλάτε προς το μικρόφωνο προς τα αριστερά σας και τώρα κάτι που θα σας εκπλήξει. Ο Ρότζερ Μπράουν, ο υπάλληλο της Επιτροπής, έχει υπηρετήσει πολύ καιρό και ενώ νόμιζε ότι είναι πολύ νεότερος, τώρα αποφάσισε να βγει στη σύνταξη, οπότε δεν μπορούμε παρά να του ευχηθούμε ε, πρώτα πρώτα τον ευχαριστούμε βέβαια, να το ευχηθούμε και καλή συνέχεια, καλή σύνταξη. Και πρόκειται και εγγράφος με επιστολή να το εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας. Πάμε τώρα στο σημείο παριθμών 3 της Μέσας Διάταξης, έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. 11 και 12 Απριλίου. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, θεωρούμε εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ακόμα μία σύντομη ανακοίνωση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Πέντε συνάδελφοι μετέβησαν στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά και στο Κόσοβο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η αποστολή. Δραστηριοποιηθήκαμε εκεί, δουλέψαμε πολύ. Ε, πήγαμε στα σύνορα με λεωφορείο και περάσαμε τα σύνορα από τη μια χώρα στην άλλη με τα πόδια διασύναμε τα σύνορα και μας περιμένει ένα άλλο λεωφορείο για να συνεχίσουμε. Έτσι μας είχαν πει. Όμως, αφού διασχίσαν το σύνορα με τα πόδια, διαπιστώσαμε ότι λεωφορείο δεν υπήρχε. Οπότε επικράτησε κάποιος μικρός πανικός. Ξαφνικά, επομένως, γραμματής και πέντε βουλευτές χαθήκανε. Ε, τελικά, πάντως, βρήκαμε ένα τοπικό λεωφορείο, ένα κτέλ, το οποίο μάλιστα ήταν και πιο φθηνό από το Πούλμαν. Οπότε να, τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε λοιπόν και τους συνεργάτες μας, βοήθησαν να είναι τόσο πετυχημένη αυτή η αποστολή και θα συνταχθεί μια έκθεση σε σχέση με τα όσα κάναμε στην αποστολή. Έχουμε δύο εκθέσεις σήμερα να εξετάσουμε. Πρώτα πρώτα για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και για το μέλλον. Έχουμε τις πράσινες βίβλους αλλά κατά τρίτον έχουμε και μια μελέτη με τίτλο «Πώς καταχράτε το οργανωμένο έγκλημα του σπόρου της ΕΕ». Ο ομιλών είναι ο εισηγητής για την πρώτη έκθεση. αλλά έχω αναλάβει και την επόμενη έκθεση, το μέλλον του ΦΠΑ. Για να δούμε τι λένε οι σημειώσει. Το 4. Είμαι εισηγητή. Συνέθηκα με την Χάιντι από την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Συνεργαστήκαμε για αυτήν την ε, έκθεση που καταλαβαίνει μόλις μία σελίδα. Έχουμε αυτές τις ε, έξι προτάσεις που είναι το πρώτο σχέδιο κειμένου. Αν εγκριθούν σήμερα θα ψηφιστεί τον Ιούλιο. Επομένως μελέτησα την πράσινη βίβλο και μπορείτε να διαπιστώσετε σε λίγο όταν δείτε αυτή την μελέτη για το οργανωμένο έγκλημα τι προβλέπετε. Ότι δηλαδή έχουμε κάποια θέματα δημοσίων συμβάσεων τα οποία επίσης εκεί αναφέρονται γιατί και εκεί αναπτύσσουν δράση αυτοί οι εγκληματίες ούτως ώστε να ξεπλύνουν χρήμα χρησιμοποιώντας τα παραθυράγια του νόμου. Το Ελληνικό Συνέδριο συνηθίσει σε έκθεση, αλλά και σε άλλες εκθέσεις, έχει πει ρητά ότι η μη τήρηση των κανόνων της δημόσιας συμβάσεις οδηγεί σαν μεγάλο ποσοστό, 43% των σφαλμάτων. Τρία τέταρτα, δηλαδή, των μετρήσιμων σφαλμάτων όσον αφορά τη συνοχή. Μεγάλο πρόβλημα, επομένω. Έχουν και σε ψηφιακή μορφή την ε, δική μας έκθεση. Και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα λάβετε το κείμενο. Οπότε, πρώτον, εδώ αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, προτρέπουμε την Επιτροπή χωρίς κάθε στέρηση να θεσπίσει κατάλληλους κανόνες για πρόληψη διαφοράς και, διαφθοράς και ευνοιοκρατίας γιατί χρειάζεται ένας κοινό ορισμός σε σχέση με το τι σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων. Να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι χρειάζεται, τόσο ώστε να φρενάρει την διαφθορά. Επίσης, προτρέπουμε την Επιτροπή να κινητοποιηθεί όσον αφορά τη διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις με διάφορες δράσεις. Χρειάζονται επίσης κάποιοι κανόνες ξεκάθαροι όσον αφορά τους καταγγέλλοντες Και παραπέμπω εδώ σε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί εκεί υπάρχουν κάποιες αξιόλογες διατάξεις που μπορούν να μας διδάξουν κάποια πράγματα. Επίσης, Κάτι άλλο πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι να ενημερώσει. Μετά την προηγούμενη Ολομέλεια, σταμάτησα στο Λουξεμβούργο, ενώ γύριζα στις Βρυξέλλες και πήγα και είδα κάποιους ε, στο ελεγκτικό συνέδριο. μισή ώρες τα λέγαμε για αυτό το θέμα. Και το ελληνικό συνέδριο διαπίστωσε ότι τα σφάλματα που προκύπτουν οφείλονται στο ότι υπάρχει άγνοια γύρω από τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Τέταρτη πρότασή μου. Και τα κρατη εκτός από την Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν σημασία στην εκπαίδευση για τους ευρωμοσταίους κανόνες. Για να είναι ενημερωμένος ο κόσμος όσοι ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις. Πέμπτη πρότασή μου. να προωθηθούν δημόσιες συμβάσεις βιώσιμου χαρακτήρα. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες που λένε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά το δίκαιο εμπόριο, το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική. Αυτά είναι κριτήρια που να διέπουν τις συμβάσεις. Όλα αυτά φαίνονται σωστά και όλα αυτά συνάδουν προς την πολιτική γενικότερα της Ένωσης. Όμως θα πρέπει όλα αυτά να είναι ξεκάθαρα. και να αποφύγουμε έτσι την απάτη. Έκτη πρόταση. Καλούμε την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα εφιστάμενα ποιοτικά κριτήρια επιλογής. να εξετάζεται η κατάσταση ταμιακών ροών κλπ. των εμπλεκομένων. Και ακριβώ τονίζω ότι η καταστάση των ροών είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, το οποίο το τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι έχει δίκιο. Και για να μπορούμε να έχουμε ποιοτικά κριτήρια χρειαζόμαστε και τις εκθέσεις και καταστάσεις ταμιακών ροών και τα δύο. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε μια υποπτία της χρηματοπιστωτικής κατάστασης του φορέα, όποιου τέλος πάντων εμπλέκεται στις συμβάσεις. Αυτά σαν ένα σχέδιο κειμένο, μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης. Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Βεβαίως και ε, το κείμενο αυτό θα το διευρύνουμε, το συζητήσουμε σήμερα και αύριο. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Η Τάλα που είναι ο σκιώδης Ευχαριστώ. Σημερίζομαι τις προτάσεις και τα σημαντικά σχόλια. Κάτι που θέλω να συμπεριληφθεί και να τονιστεί είναι ότι στις ε, δημόσιες συμβάσεις πρέπει να πλουστευτούν οι διαδικασίες για να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκείνες που απασχολούν τους περισσότερους στην Ευρώπη. Και καμιά φορά οι διαδικασίες αυτές είναι υπερβολικά δύσκολες για αυτές. Να επικεντρωθούμε εκεί λοιπόν, να πλουστεύσουμε τη διαδικασία που έχουν να αντιμετωπίσουν, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ωφεληθούν. Τώρα οι δημόσιες συμβάσεις, η ευρωπαϊκή χρήση τους πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και στα πλαίσια της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 υπάρχουν κάποιοι στόχοι εκεί όπως ποσοστό απασχόλησης ή θέματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Υπάρχουν ε, δημόσιες συμβάσεις που μπορούν στρατηγικά να αξιοποιηθούν από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη καλό είναι να σκεφτούν πώς θα γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Αυτές είναι κάποιες ιδέες που ίσως πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα των δημοσίων συμβάσεων, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούμε από εκεί να χάσουμε δισεκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι κάθε, χρώμα, κάθε χώρα ποσοστία χάνει αντίστοιχο το ίδιο ποσοστό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είμαι πεπισμένο ότι πρέπει σήμερα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη ότι κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, έχει διαφορετική ιστορία και καταλαβαίνει διαφορετικά το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Η Επιτροπή μας έχει την αποστολή να ελέγξει τι προβλήματα υπάρχουν στις διάφορες ε, χώρες. Όπως είπατε, θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν κάποια σημεία επαφής και πιστεύω ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αρχίσουν να συνεργάζονται με αυτά τα σημεία επαφή για να καταλάβουν τι διαφορέ που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν δυσκολίε με αυτέ τι διαδικασίε και σε μερικέ περιπτώσει δεν μπορούν καν να συμμετάσχουν στι δημόσιε συμβάσει. Γιατί είναι πολύ περίπλοκε οι διαδικασίες ε, για αυτέ. Ε, στην περίπτωση τη Λιθουανίας, ας πούμε, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από το 2004 ένα συγκεκριμένο μοντέλο ένα μοντέλο το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε και μπορούμε να προοδεύσουμε στο σύστημά μας ε, των δημοσίων συμβάσεων. Όχι μόνο εμείς στη Λιθουανία, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, το ηλεκτρονικό, η ηλεκτρονική πλευρά των συμβάσεων είναι πολύ σημαντική. Η επιμελητία σε κάθε χώρα κάθε χώρα πρέπει να δημιουργήσει συγκεκριμένη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Εμείς στη Λιθουανία έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα όπου ε, δίνουμε κάποια προνόμια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Ε, συνεργαζόμαστε ακόμη και με τα συνδικάτα σε αυτόν τον τομέα και ορισμένες αρχές πραγματικά είναι χρήσιμες για να προωθήσουμε το σύστημά μας. Ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς Θέλουν όμως να κρατήσουν το παλιό σύστημα. Και έτσι δημιουργούνται προβλήματα. Γενικά, είμαι ευγνώμων προς τον συνάδελφό μου που μίλησε για τη δημιουργία συγκεκριμένων αρχών. Ελπίζω στο μέλλον να δημιουργήσουμε καλύτερο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και να εξασφαλίσουμε ψηλή ποιότητα. Ξέρω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ακόμα πολλά κράτη-μέλη που πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να βελτιώσουν το σύστημά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί στα διάφορα κράτη-μέλη και να θεσπίσει τι αρχέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι δημόσιε συμβάσει που δεν θα αφορούν την ειδική κατάσταση του κάθε κράτου μέλου, θα είναι αρχέ που ισχύουν γενικά. Ευχαριστώ, κυρία Αρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Τρία σχόλια για τα συμπεράσματά σας. Λέτε ότι οι δημόσιες ε, συμβάσεις και οι κανόνες ε, είναι υπεύθυνοι για το 43% όλων των ε, λαθών. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει πει ποιο είναι το πρόβλημα, έλλειψη αφήνειας των κανόνων, πολιτιστικά προβλήματα στα διάφορα κράτη-μέλη που επηρεάζουν τον τρόπο που εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες. Για το συμπέρασμα συμπαριθμών 3. Μιλάτε για την προστασία εκείνων που λένε ποιο είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα η Κομισιόν θα πρέπει να έχει, να έχει συγκεκριμένους κανόνες για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Μία, ένα μήνα πριν ε, κάναμε μία μελέτη. Ε, δεν είχαμε και τότε πολλούς ευρωβουλευτές. Δεν νομίζουμε ότι προστατεύουμε αρκετά αυτά τα άτομα τα οποία μιλάνε ανοιχτά για το πρόβλημα. Περιμένετε πολλά, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυτόν τον τομέα, στην προστασία αυτών των ανθρώπων ακόμη πιο σημαντικό, στο σημείο 6 ζητάτε να αντικαταστήσουμε τους ισολογισμούς με δηλώσεις ε, για την ταμιακή κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε τους ε, ισολογισμούς αυτούς. Δεν πρέπει να τους εγκαταλείψουμε. Γιατί αυτό είναι το νομικό έγγραφο πάνω στο οποίο βασιζόμαστε. Και πάνω εκεί βασίζουμε τις αξιολογήσεις μας όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με την Ελλάδα μας οδηγούν σε ένα σκεπτικισμό για τους ισολογισμούς βέβαια. Αλλά ο ισολογισμός είναι το πιο σημαντικό έγγραφο και με βάση του, τον ισολογισμό φτιάχνουμε τους δείκτες, προσμετρώμε τους δείκτες. Άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την έκθεση. Αργότερα θα συζητήσουμε για το οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα στα πλαίσια που συζητάμε και το ανέφερε ο εισηγητής επίσης στο σημείο 3. Λέει ότι είναι σημαντικό να προληφθεί η διαφθορά. Όταν μιλάμε για διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα που πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε. Πρώτον, καμιά φορά υπάρχει μια προσφορά η οποία ε, προσαρμόζεται ειδικά για να προτιμηθεί. Και η διαδικασία δεν είναι απόλυτα ε, διαφανής. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν οι δημόσιοι ανοιχτοί διαγωνισμοί γίνονται για να ξεπληθεί χρήμα. Καμιά φορά η εταιρεία κάνει πολύ χαμηλή προσφορά που φαίνεται καλή στο έγγραφο, αλλά πίσω κρύβεται μια πρόθεση ξεπλήματος χρήματος. Πήγαμε στην Ιταλία βέβαια, είδαμε την κατάσταση μετά το σεισμό στην Λάκουλα όπου έπρεπε να γίνουν δημόσιες προσφορές για την ανασυγκρότηση, ανοικοδόμηση της περιοχής. Υπήρχαν έξι που έκαναν και 1.500 υπεργολάβοι και πάνω από το 20% αυτών των 1.500 δεν μπορούσαν να τεκμηριώσουν ότι δεν είχαν δεσμούς με την μαφία, άρα δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα κριτήρια. Μια τέτοια περίπτωση ε, εμείς πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι έχουμε δύο επίπεδα στη διαφθορά εδώ. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητήσουμε το σημείο 3. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στρέφομαι προς την Κομισιόν. Μήπως θέλει κάποιος να πει κάτι. Κομισιόν. Μάλιστα, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν άνοιξε αυτή τη γενική συζήτηση για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και όλα τα θέματα που αναφέρεται στην έκθεσή σας αποτελούν αντικείμενο ευρέως προβληματισμού. Είχαμε ένα σημαντικό αριθμό απαντήσεων που ελάβαμε ε, ε, στη, για την ε, Πράσινη Βίβλο επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν τα θέματα που εγείρατε κι εσείς στην έκθεσή σας. Μπορούμε να πούμε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις στα πλαίσια του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις ε, αυτές θα, λάβουν, θα κατατεθούν ως επιτοπλίστων ε, κατά το τέλος του έτους και ουσιαστικά ο άλλος πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι η αξιολόγηση που διεξάγεται για την ε, για το προηγούμενο, το τωρινό δηλαδή νομοθετικό πλαίσιο, που και αυτό θα εξεταστεί από την Κομισιόν για να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις ε, για το νέο νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ανδρέασεν. Κάνατε μία ερώτηση για το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με το ποσοστό των σφαλμάτων. Ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού, α, είδα ότι συζητούσατε, να, να περιμένω. Η κυρία Ανδρέασεν έκανε μία ερώτηση ε, προς το ελεγκτικό συνέδριο για το ποσοστό των σφαλμάτων και αν ε, έχουν ας πούμε επηρεαστεί πολιτισμικά από χώρα σε χώρα. Ίσως μπορείτε αργότερα να απαντήσετε στην κυρία Ανδρέασεν, αν δεν θέλετε τώρα. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε τώρα. Αλλά σημειώσαμε το ερώτημα της κυρίας Ανδρέασεν και θα επανέλθουμε και θα τις απαντήσουμε. Δημερός όμως. Εντάξει, δεν ζητεί άλλο το λόγο. Οπότε, ω ε, εισηγητή, ε, θα προσπαθήσω να σχολιάσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο. Ναι, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούσαμε έναν αριθμό από σχόλια, ότι οι διαδικασίες δηλαδή θα πρέπει να είναι λιγότερο διοικητικά επαχθείς. Το ξέρω αυτό και προτίθεμε να προσθέσω μια τροπολογία μετά από διαβουλεύσεις με τους συναδέλφους να καταλήξουμε σε ένα κείμενο από κοινού. Ένα σημαντικό τομέα εδώ είναι ότι θα πρέπει ίσως να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να είναι ας πούμε σαν διαβατήριο. Τι θα είναι δηλαδή αυτό. Οι επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, οι ΜΜΕ, θα υποβάλουν ένα φάκελο άπαξ που θα περιγράφει τη θέση τους, ε, την κατάστασή τους, που δραστηριοποιούνται, τι ε, στόχους έχουν, θα επιθεωρηθούν άπαξ, θα πάρουν το διαβατήριό τους και με αυτό το διαβατήριο θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασία δημοσίων συμβάσεων χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να τα ξαναλένε από την αρχή. Γιατί καμιά φορά συμμετέχουν 10 ή 15 φορές σε κάποια διαδικασία δημοσίων συμβάσεων. Δεν θα χρειάζεται λοιπόν να ξανακάνουν αυτή τη διαδικασία τη διοικητική 15 φορές. Θα έχουν, ε, τους χορηγείται άπαξ ένα διαβατήριο και αν κερδίζουν ένα διαγωνισμό θα ελέγχουμε βέβαια αν πληρούν τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο διαβατήριο. Αυτός θα είναι ένας τρόπος να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κοιτάξω να γράψω ένα κείμενο και θα το στείλω και στους συναδέλφους που είναι εδώ για να δούμε αν συμφωνείτε. Για το αν μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια κοινή τροπολογία για τις μιμίες. Τώρα, η ερώτηση για το τελευταίο σημείο της κυρίας Ανδρέασεν, τις ε, ετήσιες εκθέσεις ε, και τις δηλώσεις για την ταμιακή κατάσταση. Ίσως δεν τα είπα ε, αρκετά καθαρά. Είπα στην αρχή ότι έκανα ένα λάθος στην αρχή της διαδικασίας. Νομίζω, όπως και εσείς ε, είπατε πολύ σωστά, ότι χρειάζεται η ετήσια έκθεση και οι καταστάσεις ταμιακών ροών. Και τα δύο χρειάζονται. Οπότε δεν θα υπερτερεί μία της, ε, της άλλης, θα αποτελούν κομμάτι της ίδιας προσέγγισης. Τώρα, αυτοί που προβαίνουν σε αποκαλύψεις. Ναι, πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι εδώ. Είχαμε την, τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Κομισιόν δεν απάντησε ευθέως αν καλύπτεται ή αν θέλει να κάνει κάτι. Θα το δούμε διμερώς. Η πρόταση πάντως νομίζω ότι είναι καλή. Ο κύριος Σόντεργαρντ έκανε μια ανάλυση για το οικονομικό έγκλημα. Θα ακούσουμε περισσότερα όταν πάμε να παρουσιάσουμε τη σχετική έκθεση. Αν υπάρχει κάποια πρόταση για τροπολογία πάνω σε αυτό το θέμα, ευχαρίστω να την ε, δεχτούμε γιατί θα είναι πολύ καλή. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, κλείνουμε προς το παρόν το ζήτημα αυτό, το σημείο αυτό για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 23η Ιουνίου, η επόμενη Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφιστεί μετά στην Κοκομπού στη συνεδρίαση 13 και 14 Ιουλίου. Θα πάει μετά στην Ίμκο για να ληφθεί υπόψη δηλαδή, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην συνεδρίασή του στις 19 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια θα περάσει μετά, και θα περάσει μετά στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Αυτό είναι το πλάνο μας. Κλείνουμε λοιπόν προς ώρας και πάμε στο σημείο 5. Ε, είναι λίγο one man show ε, σήμερα η κατάσταση. Πάλι εγώ είμαι ο εισηγητής, ε, ο συντάκτης της γνωμοδότησης μάλλον για την Πράσινη Βίβλο και το μέλλον του ΦΠΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η απάτη στο επίπεδο του ΦΠΑ είναι μια πολύ σημαντική μορφή απάτης και εγκληματικότητας και δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το θέμα αυτό εδώ, στην Κοκομπή. Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να κλέψει κανείς σημαντικά ποσά. να, τα κλέψει αυτά τα ποσά από τα κρατικά ταμεία αλλά και από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στη μελέτη που θα σας παρουσιάσουμε ε, και που έχει γίνει υπό την αιγίδα του κυρίου Σόντεργαρτ, μιλάμε ακριβώς για αυτό το πρόβλημα. Σε αυτή τη μελέτη υπάρχει και ένα κεφάλαιο που αφορά και το καρουσέλ, ε, την απάτη αυτή ε, για το ΦΠΑ, στο 3-5. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αυτό το θέμα. Το 2007 υπήρχε μια συγκεκριμένη έκθεση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Επίσης και το 2007 το προηγούμενο κοινοβούλιο εξέτασε αυτό το θέμα και μάλιστα εγώ ήμουν ο συντάκτης αυτής της έκθεσης. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2008 υιοθετήθηκε η έκθεση αυτή και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρή μορφή εγκληματικότητα ασχολούμαστε με αυτό. Είναι πολύ εύκολο να βρει κανεί πολλά, πολλά ποσά, μεγάλα ποσά. Τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Μιλάμε για 200 με 500 δισεκατομμύρια ευρώ. και ε, συνολικά είναι τα ποσά αυτά της απάτης και τα ποσά απάτης του ΦΠΑ 100 δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2005-2006, 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν, ε, κλάπησαν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα και θα πρέπει να το παρατηρήσουμε. Ε, έχω δέκα συστάσεις. Μια γνωμοδότηση δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με, όλα τα, με όλες τις πτυχές ενός προβλήματος. Θα πρέπει μέσω τροπολογιών και να φτάσουμε σε ένα κείμενο πιο ισορροπημένο τελικά. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, έχω κάνει 10 συστάσεις η πρώτη σύσταση είναι μια διαπίστωση. Λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ΦΠΑ ολοκληρωμένο και επαρκώς ανθεκτικό. Εάν δεν έχουμε ένα σύστημα επαρκώς ανθεκτικό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να είναι το σημείο φετηρίας μας στη συζήτηση αυτή. Εν συνεχεία, στο δεύτερο σημείο μου, λέω ότι η απάτη αυτή με το ΦΠΑ είναι διασυνοριακή και επομένως θα πρέπει να έχουμε και διασυνοριακή δίωξη. Και αυτό τι σημαίνει έντονη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Όταν ετοίμασα την προηγούμενη εκθεσή μου του 2008, αλλά και όταν ετοίμασα αυτή τη γνωμοδότηση, συζήτησα με επιθεωρητές από τις διάφορες φορολογικές υπηρεσίε και όταν ακούμε αυτά τα άτομα μαθαίνετε απίστευτα πράγματα. Ε, πραγματικά πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα. Ε, στην σύσταση παριθμών 3 μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρη ορισμό στο κοινοτικό δίκαιο για αυτά τα, αυτές τις απάτες τύπου καρουσέλ εναντίον του ΦΠΑ που είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη η μορφή απάτη. Επίση λέω ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε τι διοικητικέ ποινέ και κυρώσει. Αυτό είναι εκ των όνου για να έχουμε ένα σύστημα και να κάνουμε διασυνοριακές έρευνε. Θα πρέπει να διώκουμε αυτή την απάτη. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ε, αυτό το πρόβλημα, οι επιθεωρητές δηλαδή, ε, μας λένε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η εναρμόνιση για να μπορέσουν να δουλέψουν αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Τέταρτη σύσταση, εν συνεχεία. Χρειάζεται ένα συντονισμό ε, πιο έντονο και πιο ταχύ μεταξύ των κρατών μελών. Χρειάζονται πιο άμεσε επαφέ μεταξύ των τοπικών φορολογικών υπηρεσιών και μεταξύ των ε, διαφόρων υπηρεσιών που κάνουν τις ε, επιθεωρήσεις. Οι αρμόδιοι μου λένε ότι συχνά παίρνουν πρωτοβουλία για να προσπαθήσουν να συνεργαστούν και προσπαθήσουν, προσπαθούν να συνεργαστούν. Υπάρχουν συνεδριάσεις μέσω του φυσκάλης, μπορεί ο κάθε επιθεωρητής από μια χώρα να έρθει σε επαφή ας πούμε, με τους Ιταλούς, Λιθουανούς, Μαλτέζους ομόλογους, ομόλογους τους για να μάθουν πράγματα, για να δουν τι αντιμετωπίζουν εκείνοι, τι εμπειρία έχουν οι συνάδελφοί τους από άλλες χώρες. Και χάρη σε αυτή την ε, εμπειρία ανοίγουν και τα μάτια τους για αυτές τις απάτες, ας πούμε τις απάτες τύπου καρουσέλα. Αλλά αυτά θα πρέπει να γίνονται και με επίσημο τρόπο, όχι μόνο ανεπίσημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι εκ των όνου κάνευ αυτός ο συντονισμός να πλαισιώνεται καλύτερα. Επίσης, θα πρέπει η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται με πιο σωστό τρόπο, πιο πλαισιωμένο, γιατί η αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών μελών είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στο σημείο 7 θα πρέπει η νομοθεσία να απλουστευτεί, να παγιωθεί, να ενοποιηθεί, να δούμε τα αδύναμα σημεία του συστήματος. Έχει γίνει βέβαια μια προσπάθεια εν μέρη, αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε και να καλύψουμε όλα τα παραθυράκια. Όχι μόνο να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη με την Κομισιόν, αλλά να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Θα πρέπει να έχουν το κίνητρο για να συνεργαστούν. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όταν ετοίμασα την έκθεση που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου του 2008, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που είναι πολύ διστακτικά ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους μόνα τους. Εν συνεχεία, θα πρέπει η νομοθεσία για το ΦΠΑ, και αυτό είναι και το αντικείμενο του της πράσινης βίβλου της Κομισιόν να απλουστευτεί και να ενοποιηθεί. Κάτι τώρα που μου λένε οι αρμόδιοι επαγγελματίε, οι επιθεωρητές δηλαδή. Μου λένε ότι συχνά ξεκινάνε μία έρευνα, παραδείγματος χάρη ένας Βέλγος επιθεωρητής, θα πρέπει να ερευνήσει ένα καρουσέλ που τον οδηγεί, που στρέφει το βλέμμα του στη Γερμανία. Ε, για τον Βέλγο η Γερμανία δεν είναι πρόβλημα, γιατί συνήθως, συνήθως μπορεί να πάρει το, γερμανικό κείμενο και να το διαβάσει. Ε, το, τα γαλλικά τα καταλαβαίνω σχεδόν όλοι στο Βέλγιο και τα αγγλικά επίσης. Αλλά αν το καρουσέλ αφορά ας πούμε την Πολωνία, την Ουγγαρία ή την Τσεχία και αν πρέπει να συνειδητοποιήσει ο επιθεωρητής αυτός τι προβλέπει η νομοθεσία των χωρών αυτών δεν καταλαβαίνουν μου λένε οι άνθρωποι αυτοί, εγώ τι να κάνω, α πούμε. Δεν καταλαβαίνω πολωνικά, δεν καταλαβαίνω ουγγρικά, δεν καταλαβαίνω τσέχικα. Άρα δεν ξέρω τι προβλέπει η νομοθεσία. Καλό θα ήταν λοιπόν τα κράτη-μέλη να μεταφράσουν τι νομοθεσίε του για το ΦΠΑ σε κάποιε πιο κοινέ γλώσσε. Ε, εγώ πρότεινα τα αγγλικά, ε, γαλλικά και γερμανικά, που είναι και τρει γλώσσε εργασία τη Κομισιόν. Ε, ξέρω ότι όταν το πούμε αυτό, η Ισπανία αμέσω θα πηδήξουν και θα πούνε Α, Ισπανικά, Ισπανικά. Αλλά νομίζω ότι αν αυτή η νομοθεσία υπήρχε στη διάθεση όλων στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ε, οι επαγγελματίες, οι επιθεωρητές ας πούμε, θα διευκόλυναν, θα, θα βοηθούνταν πραγματικά. Εν συνεχεία, η νομοθεσία, η σύσταση μάλλον Eurofisk, είναι κάτι πολύ πρόσφατο από τον Νοέμβριο του 2010 και μάλιστα στη σύστασή μου του 2008 είχα μιλήσει για αυτό το δίκτυο. Ε, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε τώρα περισσότερο για να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με σκοπό την καταπολέμηση αυτής της απάτης. Εδώ συστήνω προς την Κομισιόν να δίνει τακτικά στο Κοινοβούλιο εκθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του δικτύου. Τουλάχιστον στην ΚΟΚΟΜΠΙ και στην ΙΜΚΟ για να βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αν πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση, αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι ή όχι. Νομίζω ότι αυτές ε, οι εκθέσεις επίσης πρέπει να δημοσιοποιούνται. 8η σύσταση. Είναι μια σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ να ενισχύσουμε το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για, την, για το ΦΠΑ, περιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για τη συγκέντρωση και καταγραφή των δεδομένων. Εγώ είδα συγκεκριμένες περιπτώσεις και είδα ότι οι εγκληματίες είναι πάρα πολύ ευρηματικοί, δουλεύουν πάρα πολύ γοργά, αλλάζουν την μέθοδό του πολύ γρήγορα, αλλάζουν τις δομές τους, εξαφανίζονται, χρησιμοποιούν ε, αχυράνθρωπου. επομένως θα πρέπει και εμείς να, συζητάμε, να, δανδρούμε πάρα πολύ ταχαίω για να αντιμετωπίσουμε την απάτη αυτή. Εν συνεχεία, δεύτερο στοιχείο, η πρόσβαση στις ε, πληροφορίες για τις ε, υπηρεσίες επιθεώρησης πιστεύ, ε, μας λένε ότι και εκεί πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Υπάρχουν και δύο τελευταίες συστάσεις. Τώρα εδώ είναι μια πιο γενική συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ΦΠΑ ε, στις επαφές που είχα με τους επαγγελματίες, με τους επιθεωρητές κτλ. Συνειδητοποίησα, από αυτές τις συζητήσεις συνειδητοποίησα ότι είναι σημαντικό να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί μας λένε ότι το σύστημα Το reverse charge, όπως λέμε στα αγγλικά, είναι ένα σύστημα που θα πρέπει να ξαναδούμε. Αυτό το μηχανισμό δηλαδή της αντίστροφης χρέωσης του ΦΠΑ. Αυτό το τσεκάραμε, το ελέγξαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το χρησιμοποιούμε για τους υπολογιστές και για τα κινητά και μου λένε ότι έδωσε καλά ε, αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στην σύστασή μου 9 στρέφαμε προς την Κομισιόν για να τη ρωτήσω αν σκοπεύει να υιοθετήσει αυτό το σύστημα. Ε, κοιτάτε τι συμβαίνει σε άλλες, άλλε άλλες χώρες. Βγάζετε συμπεράσματα. Τη ρωτώ. Και στο 10 συστήνω, προτρέπω στην Επιτροπή, να κάνει νομοθετικές προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν ε, τις περιπτώσεις απάτης ε, τύπου καρουσέλ στη ρίζα. καθιερώντα σε ενωσιακό επίπεδο το μηχανισμό αντίστροφη χρέωση του ΦΠΑ. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν ποια είναι η αντίδρασή τη. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τρόπο για να καταπολεμήσουμε την απάτη. Και αυτό είναι προ όφελο και των εμπόρων και προ όφελο των παραγωγών. Νομίζω ότι ο οπτικοακουστικός τομέας, τα τρόφιμα και τα ποτά, ε, το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, εξερτήματα, κινητά τηλέφωνα και εξαρτήματα, κλωστιφαντουργικά προϊόντα και αυτοκίνητα θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν αντίστροφης χρέωσης. Νομίζω ότι το συζητάει αυτή τη στιγμή η ΙΜΚΟ στα πλαίσια τη συζήτηση που γίνεται για την πράσινη βίβλο. Θα ήθελα λοιπόν οι συνάδελφοι να μου πούν τι γνώμη έχουν για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση και ελπίζω να ακούσω και κάτι, κάποια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο θέλει να αντιδράσει, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόεδρε, μια και δεν είμαστε και πολλοί, ας απαντήσω στα Ολλανδικά. Οι προτάσεις σας ε, είναι σε γενικές γραμμές εξαιρετικές. Μια σκέψη να εκφράσω και ε, στο Κοινοβούλιο, άλλωστε πάντα θέλαμε ένα σύστημα πιο ορατό και το 0,4% του ΦΠΑ καταβάλλεται στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ, αν πιω έναν καφέ ένα ποσοστό του ΦΠΑ που επιβάλλεται επιστρέφει στο, στην Ομοσπονδία, ένα άλλο στην πολιτεία ένα άλλο τμήμα του ΦΠΑ πάει στην κοινότητα όπου ζει κανεί. Μήπως λοιπόν αυτό είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να ισχύσει και στην Ευρώπη. Μπορεί να γίνουν όλα αυτά σχετικά εύκολα. Πώς ε, αξιοποιείται και πώς ελέγχεται η αξιοποίηση του ΦΠΑ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε καλύτερα αποτελέσματα να έχουμε με ένα τέτοιο σύστημα. Η κυρία Ανδρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι προτάσεις σας είναι θετικές. Να ρωτήσω μόνο αν προηγήθησαν διαβουλεύσεις με την Όλαφ, η οποία έχει ένα τμήμα ειδικό για την απάτη του ΦΠΑ. Οπότε ξέρει να μας συμβουλέψει σχετικά με τις αλλαγές που χρειάζονται τα συστήματα στην Ευρώπη. Μου κάνει εντύπωση πως δεν γίνεται μνήα της Όλαφ εδώ. Γιατί εκείνοι έχουν πολλές φορές καταπολεμήσει τέτοια, τέτοιες απάτες έχουν δηλαδή στοιχεία για το τι ποσοστό, σε τι ποσοστό ανέρχονται οι απάτες σε αυτό το τομέα και θα έχουν και κάποιες προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Άλλος κανείς, άλλο μέλος, πάμε στην Κομισιόν. Τι, πώς αντιδράτε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κάποιες γενικές αντιδράσεις. Η Κομισιόν γενικά συμφωνεί με τις συστάσεις που κάνετε. Κάποιες διευκρινήσεις να σας δώσω μόνο. Προς πληροφόρησή σας, η Κομισιόν έχει κάνει μία μελέτη για να ποσοτικοποιήσει την απάτη του ΦΠΑ, το κενό όπως λέμε ΦΠΑ και για το 2006 για 25 κράτη-μέλη, με βάση τον υπολογισμό που κάναμε μέσω ενός συμβούλου, είναι 107 δις ευρώ. Προσπαθούμε τώρα να επικαιροποιήσουμε αυτή τη μελέτη για να λάβουμε υπόψη μας και τα πιο πρόσφατα νούμερα, για τα πιο πρόσφατα έτη. Μετά από την έκθεση που παρουσιάσατε όμως ε, το 2008 για τη στρατηγική κατά της απάτης της Κομισιόν, πρόθεσαμε προωθήσαμε διάφορες δράσεις, την υιοθέτηση ενός κανονισμού για την διοικητική συνεργασία, που υιοθετήθηκε αυτός από τα κράτη-μέλη και θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτός ο κανονισμός ενισχύει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως δημιουργώντας ε, επίσημα πια το Eurofisk, που προηγουμένως δεν είχε νομική βάση σταθερή. Επίσης, ε, τονίζει και διευκολύνει τους ε, πολυμερείς ελέγχους, δηλαδή τους διασυνοριακούς, όπως ακριβώς το προτείνεται, βελτιώνοντας σημαντικά τις βάσεις δεδομένων, δηλαδή την άμεση πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες από τις φορολογικές υπηρεσίες, κάτι που λέτε και εσείς στις διάφορες Η Κομισιόν έχει το καθήκον να παρουσιάζει μια έκθεση για την ε, λειτουργία αυτής της διοικητικής συνεργασίας και η νομική βάση της Eurofisk βρίσκεται σε αυτό τον κανονισμό, ε, γι' αυτό η έκθεση της Κομισιόν θα αφορά και το EuroFisk. Ε, το EuroFisk, όπως είπατε, ξεκίνησε τη δράση του πρόσφατα. Χρειάστηκε λοιπόν να δημιουργήσουμε διάφορες δομές και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί σχετικά καλά. Μας εκπλήσει αυτό. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν μάλιστα με έντονο τρόπο, παρότι στην αρχή η συμμετοχή στο Eurofisc ήταν εθελοντική, δεν ήταν υποχρεωτική, αλλά σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στο Eurofisc. Για, πιο, ε, για το πιο συγκεκριμένο ερώτημα αυτό της ε, αντίστροφης ε, χρέωσης, πιστεύουμε ότι αυτό αυτός ο μηχανισμός μπορεί να ε, λύσει το πρόβλημα της απάτης του καρουσέλ σε συγκεκριμένους τομείς. Επίσης έχουμε δώσει εδώ διάφορες ε, παρεκκλήσεις ε, στα κράτη-μέλη στους τομείς που αναφέρατε. Υπάρχει μια πρόταση της οδηγίας ε, της Κομισιόν προς το Συμβούλιο, αλλά τα κράτη-μέλη δεν την έχουν ακόμα υιοθετήσει, που, προβλέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα σύστημα αντίστροφη χρέωσης σε ορισμένα προϊόντα χωρίς να ζητήσουν ιδιαίτερη παρέκκληση από την Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη όμως δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα για αυτό το κείμενο βρίσκεται ακόμα προ εξέταση το Συμβούλιο. Τώρα, για το μέλλον. Η Κομισιόν σκέφτεται να προτείνει ένα σύστημα γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση Ε, είχαμε το πρόβλημα της απάτης ε, και αν δοθεί παρέκκληση στα κράτη-μέλη, χρειαζόμαστε 9 μήνες. Ε, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα για να κατεπολεμήσουμε την απάτη. Γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει να... ένα σύστημα έγκαιρης αντίδρασης που μας επιτρέπει να κινητοποιηθούμε πολύ πιο γρήγορα σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης. Αυτά είχα να σας πω. Να μην ξεχνάτε ότι η πράσινη βίβλος αφορά κυρίως τις μελλοντικέ δράσεις και μία από αυτές τις δράσεις που προτείνονται στην πράσινη βίβλο, που θα πρέπει να συζητηθεί βέβαια, είναι ότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η συλλογή του ΦΠΑ από τα περισσότερα κράτη-μέλη γίνεται με τρόπο ε, απαρχιωμένο. Και επομένως είναι σημαντικό τα κρατημέλη να χρησιμοποιούν καλύτερα όλα τα μέσα που έχουν, δηλαδή μηχανοργανωμένα συστήματα συλλογής του ΦΠΑ. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ περισσότερο, ιδίως για τη μέθοδο, δηλαδή το θέμα της μεθόδου συλλογής των εσόδων από το ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή βασιζόμαστε το φορολογούμενο δηλαδή. Αυτός είναι ο βασικός παίχτης. Αυτός λαμβάνει το ΦΠΑ και αυτός τη δίνει στο ΦΠΑ. Σε ορισμένε περιπτώσει δεν την ε, δίνει με τη σειρά του στο, στο, κράτο και αυτή είναι η περίπτωση τη απάτη καρουσέλ. Θα πρέπει λοιπόν να το καταθέσουμε πιο υπεύθυνο. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή να τον παρακάμψουμε. Έχουμε σκεφτεί το σύστημα του split payment, χωριστή ε, πληρωμή που χρησιμοποιείται σε τρίτες χώρες. Δηλαδή το ΦΠΑ ε, καταβάλλεται κατευθείαν στη φορολογική υπηρεσία χωρί να περάσουν από το φορολογούμενο. Δεν είναι εκείνο υπεύθυνο για να καταβάλει το ΦΠΑ στο κράτο, α πούμε. Θα πρέπει ούτω ή άλλως να ενισχύσουμε και τον έλεγχο που γίνεται σε κοινοτικό επίπεδο για το ΦΠΑ. Αυτά είχα να σα πω προ το παρόν. Άλλο συνάδελφο θέλει να μιλήσει. σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για αυτά τα ενδιαφέροντα σχόλιά του. Είναι ενδιαφέρον το ότι το 2006 το ποσό της, απο... της απάτης έφτασε σε ύψος 107 δις ευρώ. Είναι περισσότερο από ό,τι νόμιζα. Δεν ήξερα αυτή τη μελέτη, δεν ήξερα αυτό το ποσό. Ενδιαφέρον αυτό που μου είπατε λοιπόν. θα, θα μπορούσατε να μας δώσετε αυτή την μελέτη, να την, έχει, δηλαδή, να την έχουν τα μέλη της κοκομπής στη διάθεσή τους. Ε, συνεχεία, η πρόταση της ε, Κομισιόν προς το Συμβούλιο για τις ε, ειδικέ παρεκκλήσει για το πώ μπορούμε να πλουστεύσουμε το σύστημα των παρεκκλήσεων. Θα, μπορούσα, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Μια διευκρίνηση, λέει η Κομισιόν. Δεν μιλάμε μόνο για την απάτη, αλλά για τις διαφορές μεταξύ της, του θεωρητικού ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να συλλεχθεί και του πραγματικού ποσού που συλλέχθη. Δηλαδή αφορά και την απάτη, αλλά αφορά και τα, τα λάθη, και αφορούσε μόνο τα 25 κρατη για το 2006. Πέντε χρόνια μετά είμαστε σήμερα. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό, αυτή η μελέτη στην ιστοσελίδα της Γενική Διεύθυνση Ταξούντ. Είναι στη διάθεση όλων λοιπόν. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, τελειώνουμε με αυτό το σημείο αυτό. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 23 Ιουνίου 2011, ώρα 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία 13 και 14 Ιουλίου στην Κοκομπή. Είπα ότι συμμετέχει και η ΙΜΚΟ στις ε, δημόσιες συμβάσεις και η Επιτροπή η ΕΚΟΝ θα ψηφίσει στις 19 Σεπτεμβρίου. Οπότε έχετε πολύ χρόνο. Έχουμε πολύ χρόνο για να επηρεάσουμε την Επιτροπή ΕΚΟΝ Οικονομικών Υποθέσεων. Πάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα. Πρόκειται για μία μελέτη η οποία, την οποία ανέθεσε η Επιτροπή μας για το πώς καταχράται το οργανωμένο έγκλημα του σπόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Βένσιγκ, ένας από τους ε, συντάκτες της μελέτης, της μελέτης είναι εδώ. Η PricewaterhouseCooper την ε, διεξήγαγε και προτείνω να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Βένσινγκ. Έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε πρόβλημα χρόνου. Πρώτη φορά έρχεστε εδώ. Καμιά φορά λειτουργούμε κάτω από χρονική πίεση. Σήμερα όμως όχι. Οπότε νιώστε άνετα από αυτή την άποψη. Για να μας τα παρουσιάσετε ωραία και να καταλάβουμε κι εμείς τι ακριβώς μας λέτε. και μετά ο κύριος Ζων Ντεγκάρντα επίσης θα πάρει το λόγο. Ο κύριος ε, Βάντσινγκ έχει πρώτος το λόγο. Είναι στα αγγλικά η μελέτη, κάποια πιο τεχνικά θα τα πω στα Ολλανδικά και έχω και κάποιες διαφάνειες που συνοδεύουν την παρουσίασή μου. Έχω μια μακρά ημερήσια διάταξη, αλλά έχουμε χρόνο να μην ε, τα ποδιαστικά, Καταρχήν να πω δύο λόγια για το σκοπό αυτής της μελέτης. Η μελέτη, ο στόχος της μελέτης ήταν να δούμε πώς ε, καταχράται το οργανωμένο έγκλημα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πόρους της Ένωσης και τι μπορούμε να κάνουμε. Πριν απαντήσω με το πώς και το τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνουμε κάποιες, ε, κάποιους ορισμούς, τι είναι το οργανωμένο έγκλημα, ποιοι είναι οι κοινοτικοί πόροι στα πλαίσια της μελέτης, τι αποτελεί κατάχρηση και αν καταχράτε το οργανωμένο έγκλημα και σε ποιο βαθμό και έκταση του πόρους της Ένωσης και τέλος με ποια μέσα και με ποιες μεθόδους. Πώς τέλος πάντων καταχράτε το οργανωμένο έγκλημα του πόρους της Ένωσης. Αφού απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, διατυπώνουμε συστάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην αυξημένη θωράκιση των ε, πόρων της Ένωσης. Τώρα, στα πλαίσια των ε, αρμοδιοτήτων που έχουμε, στηριχθήκαμε σε μελέτες και εκθέσεις από ελεύθερες πηγές Επίσης λάβαμε υπόψη μας τις πληροφορίες που λάβαμε από την Όλαφ, το ελεγκτικό συνέδριο, την Europol και την Eurojust και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι επικεντρωθήκαμε στην κατάχρηση των πόρων της Ένωσης το 2009. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι Πολλές πληροφορίες δεν ήταν άμεσα προσπελάσιμες. Έπρεπε να συμπεριλάβουμε και ε, πληροφορίες από προηγούμενα έτη για να ε, συναγάγουμε συμπεράσματα. Κάναμε μία μελέτη λοιπόν που στηρίζεται και σε μελέτη εγγράφων και σε συνεντεύξεις και δημόσιες ακροάσεις εδώ για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 22 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους κάναμε και μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων πάλι στο, εδώ στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ειδικού από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και από την Όλαφ και την Europol και από την διεθνή διαφάνεια επίσης για να αναφέρω ορισμένους. Τώρα, υπάρχουν προκαταρκτικά ευρήματα στην ε, ενδιάμεση έκθεση. Τώρα, πώς έγινε η μελέτη. Όπως είπαμε, πρώτα απ' όλα προσπαθήσαμε να ορίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Δεν θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος καθολικός ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος και για να παραθέσω τον κύριο Κρετέμ που είναι διευθυντή στην Όλαφ, το οργανωμένο έγκλημα αλλάζει συνεχώς ως φαινόμενο σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και οι ορισμοί του οργανωμένου εγκλήματος διαφέρουν ανάλογα με τη χρονική στιγμή και οι διάφοροι ορισμοί αντικατοπτρίζουν διάφορες γωνίες ε, πρίσματος για την προσέγγιση του θέματος και διάφορες σχολές δράσης. Ένα εναρμονισμένος ορισμό όμως χρησιμοποιείται από όλους τους ε, εμπλεκομένου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. και έτσι μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες πάνω σε μια ενιαία βάση. Είδαμε όμως ε, ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν, δεν χρησιμοποιούν έναν ορισμό, αν χρησιμοποιήσουν ορισμό. Σε αυτό θα επανέλθω αργότερα όταν πάω στα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Για τους σκοπούς της μελέτης συνδυάσαμε στοιχεία υπαρχόντων ε, ορισμών του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως αυτόν τον ορισμό που υπάρχει στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος το 2008. Προσθέσαμε εδώ και την πτυχή της σοβαρής ζημίας στην οικονομική ακαιρεότητα και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ορισμός μας και τα ιδρύματα της Ένωσης. Έτσι λοιπόν ο ορισμός μας είναι ότι είναι μια δομημένη ένωση η οποία έχει δημιουργηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και σκοπό έχει να διαπράττει αδικήματα για παράνομο προσπορισμό που προκαλούν σοβαρή βλάβη στην οικονομική δημοσιονομική ακαιρεότητα ε, και τα θεμέλια αλλά και τα ιδρύματα, τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσαμε επίσης ε, να ορίσουμε για το σκοπό της μελέτης ε, τι είναι η πόρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη μελέτη προσέχουμε ιδιαίτερα τα, τους δαπανόμενους πόρους από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους ε, ίδιους πόρους. Ε, ποσοστό του ΦΠΑ είναι εδώ και οι ειδικοί φόροι που εισπράττονται στα κράτη-μέλη θα μπορούσαν και αυτοί να θεωρηθούν ε, πόροι της Ένωσης αφού χρηματοδοτούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και επειδή ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι προσελκύουν πολλούς εγκληματίες και η κατάχρησή τους για τους σκοπούς της μελέτης, η κατάχρηση των ε, πόρων ελήφθη υπόψη και οι απάτες σε αυτό το τομέα, λαθρεμπόριο τσιγάρων για παράδειγμα κλπ. Επειδή η κατάχρηση θεωρείται κακή η εσφαλμένη χρήση, κακή χρήση, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την ε, αθέλητα λανθασμένη χρήση. Μεταξύ σκόπιμης και μη σκόπιμης χρήσης θα πρέπει να δούμε ένα, και να δούμε το εφιστάμενο ε, νομικό πλαίσιο. Εδώ η κατάχρηση θεωρείται απάτη με τους κοινοτικούς πόρους. δηλαδή ε, παραβίαση, κατάχρηση εμπιστοσύνη ε, για ε, παράνομο προσπορισμό, αθέμητο, πλεονέκτημα, όλα αυτά είναι σκόπιμες πράξεις νομική βάση για δράση σε νοσιακό επίπεδο για να ε, προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να καταπολεμήσουμε την απάτη και εδώ η σχέση ε, με την ε, έννοια απάτη στηρίζεται στο άρθρο 35 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης. Η διαχείριση και ο έλεγχος των νοσιακών πόρων ε, στηρίζονται σε μια δομή ελέγχου που περιγράφεται εκτενώς στη μελέτη μας. Ε, μια δομή ελέγχου για όλα τα κονδύλια, του σπόρους που δαπανώνται, που είναι σε διάφορες βαθμίδες ε, και πρωταρχικά η ευθύνη για αυτή τη δομή βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Σε αυτήν την δομή ελέγχου μεγάλη προσοχή αποδίδεται σε προτάσεις για έργα, ε, στις προδιαγραφές ε, των ε, διαγωνιζομένων, την ορθή οικονομική διαχείριση και γίνεται γενικός έλεγχος των διαγωνιζομένων, τις οργανώσεις που κρύβονται από πίσω, άλλοι που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και επίσης βλέπουμε και τα κέρδη που αποκομίζουν. Οι δαπάνες ε, λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη και το σύστημα ελέγχου ε, επηρεάζεται πολύ από την προσοχή που αποδίδεται σε αυτό στο επίπεδο των κρατών μελών. Επανεξέταση, εσωτερικός έλεγχος δαπανών πόρων της Ένωσης στα κράτη-μέλη γίνεται από ε, εθνικούς αξιωματούχους σε εθνικό επίπεδο και δεν γίνεται έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ή έλεγχος από ομοτήμους. ομοτήμους. Επίσης, ε, τα πρότυπα που ισχύουν για τους αξιωματούχους που κάνουν τον έλεγχο στα κράτη-μέλη διαφέρουν και μικρές διαφορές μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές στο... στην έκβαση του ελέγχου λογιστικών εσωτερικών ελέγχων κλπ. σε επίπεδο κρατών μελών. Οπότε εδώ το σύστημα επιδέχεται βελτιώσεων, πιστεύουμε. Εις ό,τι αφορά τώρα το εύρος της κατάχρησης ε, των ε, πόρων της Ένωσης ε, από το οργανωμένο έγκλημα, εδώ δεν έχουμε σχεδόν καθόλου αξιόπιστες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς Europol, Olaf ή το ελεγκτικό συνέδριο δεν ε, ήταν σε θέση, δεν μπορούσαν να μας δώσουν ξεκάθαρα στοιχεία και νούμερα. Μόνο η Europol μπόρεσε να συμβάλλει στη μελέτη με τρία περιστατικά από το 2009 και παρουσίασαν και κάποιες ε, υποθέσεις με τον ΦΠΑ, αλλά η τάξη μεγέθους της απάτης δεν μας δόθηκε. Από την άλλη πλευρά, Μας δώσανε κάποιες εκτιμήσεις η Όλαφ και η Europol δηλαδή. Η Όλαφ ανέφερε για παράδειγμα ότι το 2009-2010 σε αυτή την ετήσια έκθεση είδαν αυξανόμενες αποδείξεις ότι σε πολλές περιπτώσεις οι απάτες στα διαφορετικά ταμεία της Ένωσης είναι οργανωμένα και σχεδιασμένα και δεν ε, ε, έγιναν τυχαία, δηλαδή δεν ήταν ευκαιριακά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει την ύπαρξη κάποιας δράσης οργανωμένου εγκλήματος, αν και δεν μας δώσανε τα υποκείμενα μεγέθη. Η Europol αναφέρει ότι η απάτη στον ΦΠΑ και η απάτη στις δημόσιες συμβάσεις ε, δεν αναφέρει όμως πώς μεγάλη είναι η απάτη με τον ΦΠΑ και τις δημόσιες συμβάσεις. Τι έκταση έχουν. Ούτε δίνει λεπτομέρ... δεν δίνουν ε, λεπτομέρειες για τις δηλώσεις που έκαναν σε μας. Οπότε για να απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με το πώς καταχρώνται τους πόρους οι εργομένοι εγκληματίες, οι πηγές πληροφοριών μας είναι περιορισμένες, κυρίως ανοιχτής πηγής. Αυτά που συνάπτονται εν παραρτήματι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο website σήμερα. Έχουμε ένα hard copy, αλλά τέλος πάντων θα σας παρουσιάσουμε την τελική εκδοχή, το κειμένο και έχουμε επομένω αυτό το κατάλογο με πολλές, αρκετές περιπτώσεις Ανοιχτή πηγή που θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρη περίπτωση απάντηση που αφορά του κοινοτικού πόρου. Όμω, δεν έχουμε λάβει κάποια επαληθευμένα στοιχεία από τα θεσμικά όργανα και τι περιφερειακές υπηρεσίες, μόνο από την Eurojust κάποιες, ε, φακέλου υποθέσεων, από την Όλαφ κάποιες αναλύσεις ε, του πρόσφατου παρελθόντος και Από τη Europol δεν πήραμε τίποτε το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πολύ ή από το ε, συνέδριο. Οπότε, γι' αυτό και μπορούμε μόνο να συναγάγουμε κάποια γενικού χαρακτήρα συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να ανασχέσουμε αυτό το κύμα ρωμένου εγκλήματος στην Ένωση. Είναι αυτά τα οποία στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να δείτε. Οπότε και έχουμε κάποιου είδου γενικά χαρακτηριστικά του, του, του, των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι έχουμε πάνω από δύο φυσικά πρόσωπα ή και εταιρείε που εμπλέκονται και ότι τα περισσότερα εγκληματικά δίκτυα ε, έχουν διεθνή δράση. Τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δεν θα σας εκπλήξει ότι είναι η δωροδοκία, η διαφθορά, Ε, πλαστογραφία, παραποίηση εγγράφων, πιστοποιητικών, ε, περί τα επιδόματα απάτη, ε, παράκαμψη των ε, διαδικασιών, τα παθράκια στον νόμο δηλαδή, καθώς και επίσης και εικονικές εταιρείες. Επίσης, προσέζει, πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, ούτως ώστε να προστατευτεί το οικονομικό συμφέρον, τα οικονομικά συμφέροντα τέλο πάντων τη ε, Ένωση. Και αναφέρει το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε ε, προκλήσει σε αυτέ τι ανακοινώσει τη και ε, τι πρωτοβουλίε. Πρώτα-πρώτα, πώ θα ξεπεράσουν τι δυσκολίε όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων για το βαθμό που λαμβάνει η χώρα η απάτη, αλλά και η ποινική δίωξη, η πραγματική σε δικαστήριο, τι γίνεται με τι διασυνοριακές ε, περιπτώσει, πώ μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικά δικαστήρια όσον αφορά τι ποινικέ δίκες. Να, ε, κάποιε από αυτέ τι πρόσφατε ε, δηλώσει κλπ. όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφωνών τη Ένωση. Επίση, έχει προταθεί η μεταρρύθμιση τη Όλαφ, πολέμηση της διαφθοράς και επίσης διαβούλευση όσον αφορά τον εξυγχρονισμό τη πολιτική για τι δημόσιε συμβάσει. Οπότε μπορούμε να διαπιστώσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες τα εξή. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρει το οργανωμένο έγκλημα ή τέλο πάντων δεν εστιάζει εκεί την προσοχή του ενδιαφέροντε μόνο εκεί. Ε, διότι από αυτές τις πρωτοβουλίες προκύπτει ότι η τελο παντων δεν εστιαζει εκει την προσοχη του ενδιαφεροντες μονο εκει ε διοτι απο αυτες τις πρωτοβουλιες προκυπτει οτι η δραση της Κομισιόν κατευθύνεται κατά οποιασδήποτε απάτης διαφθοράς πέραν της μορφής διάρθρωσης της απάτης, πέραν ε, του το αν είναι στιγμίο το αδίκημα ή διαρκές και οπότε αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κάπως τυχαία προσέγγιση ε, γιατί πάρα πολλές φορές δυσκολεύεται στο να βρει ακριβή δεδομένα και στοιχεία για τον βαθμό ε, της απάτης την τάξη μεγέθου. Ε, δεν υπάρχουν μηχανισμοί αξιολόγηση, Επομένω χρειάζονται και καλύτερα στατιστικά κοινοτικά. Οπότε και τίνουμε να συμφωνήσουμε με αυτό το τελευταίο σημείο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά αυτές τις δυσκολίες ε, απόσπασης αξιόπιστων ε, στοιχείων και αξιολόγηση. Όλα αυτά μα οδηγούν σε κάποια συμπράσματα. Πρώτα-πρώτα, χρειάζεται κάποιο είδου κοινή αισθήση τη προσοχής στο τι γίνεται για αυτό το οργανωμένο έγκλημα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα και για την απάτη και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Όμως η καταπολέμηση της κατάχρησης των χώρων από το, το, το, από οργανωμένο έγκλημα και αυτό θα πρέπει να το καλύψουν τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίε τη Ένωση. Επίσης, στα πλαίσια αυτών των ε, συμπερασμάτων διαπιστώνουμε ότι κάποια όργανα και υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν ενιαίο ορισμό του τι να πει οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό πιστεύουμε ότι αποτελεί έναν ε, φραγμό στην αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα για το θέμα και άρα είναι δύσκολο κανείς να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με το σε τι βαθμό γίνεται αυτή η κατάχρηση των κοινοτικών πόρων. Άρα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να θωρακίσουν περισσότερο τους κοινοτικούς πόρους. Επίσης υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της διαχείρισης, του οικονομικού ελέγχου, ε, της, δαπάνη δαπάνης των γενικών πόρων και στα κράτη-μέλη αλλά και στο ενωσιακό επίπεδο. Οπότε και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε την περίπτωση της απάντησης. Αυτό χρειάζεται εις όλα τα επίπεδα διαχείρισης και όχι τόσο όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματο, αλλά στο να υπάρχει επίγνωση των πιθανότητων αντικανονικών ενεργειών και απάντηση σχέση με τους πόρους και το τι μπορεί να κάνει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Επίσης, Παρακάτω. Πάμε σε κάποιες μας συστάσει. Πρώτον, έχουμε εδώ μια σειρά από τέτοιε συστάσει. όπου συστήνουμε περισσότερη εστίαση ή στην απάτη. να βρεθούν κοινοί ορισμοί αλλά και να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ενιαίος ορισμός, κοινός ορισμός και για άλλες έννοιες για το θέμα, όπως κατάχρηση, απάτη, κοινοτικός πόρος και ορισμός να χρησιμοποιείται από όλους τους εμπλεκομένους όργανα κλπ. Επίσης, κάπου να αρχιοθετούνται όλες οι υποθέσεις τέτοιων παραβάσεων και εγκλημάτων. Αυτό να γίνεται κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, Ούτως ώστε να είναι εφικτό να κάνει κανείς συγκρίσεις, να διασυνδέει υποθέσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και να μπορεί να συνδέει κανείς περιπτώσεις μεταξύ των καθέκαστων περιπτώσεων απατών, οργανωμένων εγκλήματος, αντικανονικοτήτων κλπ. Άλλη μας τώρα σύσταση είναι όλα, Europol και Eurojust, να συστρατευτούν μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο και όλοι μαζί να εστιάσουν τη δράση τους σε καταχρήσεις, σε απάτες που κάνουν εις βάρος των κοινωτικών πόρων οι οργανωμένοι κλιματίες. Και να δούμε αυτό το δύσκολο θέμα, το, το βαθμό στον οποίο εξαπατά την Ένωση το οργανωμένο έγκλημα. Άλλο να επιφέρουμε κάποια βελτίωση όσον αφορά το επίπεδο της ποιότητας του οικονομικού ελέγχου για τους οικονομικούς πόρους. Λέμε εδώ να δούμε αν είναι δυνατόν να έχουμε εσωτερικό έλεγχο τι γίνεται εάν τα λεφτά να πηγαίνουν στους επιλέξιμους στο, κράτος μέλος να, να, να, κάποιοι άλλοι ε, υπάλληλοι να τα, να τα εκτρέπουν αλλού. Καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα πανούνται τελικά αυτοί οι πόροι. Επίσης, άλλη σύσταση. να συνειδητοποιηθεί περισσότερο, να υπάρχει περισσότερη ενάργεια ούτως υπήν σε σχέση με τις απάτες και να να, να βαθμιστεί, να, να, να νιωθεί η έννοια της μηδενικής ανοχής. Να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα πάγιας, μόνιμης ανάσχεσης της απάτης. Και σε επίπεδο κρατών μελών, πάντα όσον αφορά τα κοινοτικά χρήματα. Ξεκάθαρες πολιτικές, ε, επίσης να υπάρχει ε, εξαντλητική εξέταση του προφίλ του κάθε προσλαμβανομένου. Και έτσι να έχουμε και τις προσλήψεις αλλά και τις δραστηριότητε που γίνονται από το προσωπικό κάθε φορά μέσα σε συνθήκες ασφάλειας. Επίσης λέμε ότι θα πρέπει να ερευνηθεί η δυνατότητα του να χρησιμοποιούνται κάποιο είδους εργαλεία μέσα υποστήριξης αυτού του είδους το, το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά είναι επιλέξιμοι για τα κοινωνικά χρήματα και έτσι να ανοιχνεύονται οι, οι απάτες. Κάποιο είδους εγκόλπιο νομικών μέσων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και επομένως, εάν διαπιστώνονται κίνδυνοι να αναστέλλονται οι πληρωμές να οι χρηματοδοτήσει έργων και προγραμμάτων. Επίση, κάποια άλλα μέσα, ώστε να γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου και επίσης ε, αξιολόγηση και να έχουμε και κάποιες διαδικασίες εξαίρεσης, αποκλεισμού. Επίσης να υπάρχει κάποιο είδους ε, λειτουργική δομή, να υπάρχει μια καινούρια κουλτούρα ε, όσον αφορά τις καταγγελίες, να προστατεύονται οι καταγγέλλοντες, οι whistleblowers και το ίδιο να αφορά και το προσωπικό το οποίο επισημαίνει και αναφέρει περιπτώσεις απάτης. Και σε επίπεδο ένωσης, το αρθρο 22 22α και 22β να αναθεωρηθούν, τα οποία περιέχονται στον κανονισμό λειτουργίας. Ε, επίσης και η πληροφορική να υποστηρίζει αυτές τις ενέργειες και με, με κάποιο είδους εφαρμογές λογισμικού software. Οπότε να δούμε τι άλλες στάσεις έχουμε εδώ. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει και λογοδοσία υποχρέωση λογοδοσίας και αυτό να χρήση παντό μέσου τόσο ώστε να έχουμε δημοσιοποίηση, να έχουμε διάχυση των, των σχετικών ε, πληροφοριών όσον αφορά το τι γίνεται με πόρους και έτσι να ξέρει ο κόσμος. Επίσης, λέμε και για την ε, απάτη ΦΠΑ ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη-μέλη να έχουν μία αντιστροφή τις επιβάρυνσεις όσον αφορά τις περιπτώσεις απάτης με τον ΦΠΑ. Αυτό κάπως είναι τεχνικό θέμα το οποίο το αναλύουμε στην ε, έκθεση. Εδώ θα βάζουμε τελεία στην εισήγησή μας και έχετε τη σκητάλη. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Και τώρα ο λόγος στον εισηγητή τον κύριο Σόντεργαρτ ο οποίος με τη σειρά του θα μας ε, εξηγήσει πώς βλέπει τα πράγματα. Έχετε όμως και κάποιες ερωτήσεις. Σόντεργαρτ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Είναι δύο οι βασικοί λόγοι για τους οποίους εγώ ε, εξ αρχής είχα προτείνει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα πρέπει να προβεί σε αυτή την ε, έκθεση, σε αυτή τη μελέτη σε σχέση με το τι κάνει το οργανωμένο έγκλημα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων και πόλων της Ένωσης. Και επομένως έτσι μπορούμε να συμφωνήσουμε το ότι θα πρέπει πρώτα πρώτα να προστατεύσουμε το συμφέρον του προλογούμενου. Γιατί ό,τι και να πιστεύει κανένας για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να συμφωνεί ότι η απάτη εις βάρος ε, των κοινωτικών πόρων είναι κάτι το καταστροφικό, είναι κάτι το απαράδεκτο. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει και για λόγους προστασίας της δημοκρατίας να προβούμε στις σχετικές ενέργειες. Όταν έχουμε οργανωμένο έγκλημα το οποίο είναι τόσο ισχυρό, δεν πρόκειται εδώ απλώς περί εγκλήματος ή πρόκειται περί εισδοχής διάβρωσης του πολιτικού συστήματος και της διοίκησης. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να συνεχίζεται με εγκληματική δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει δίωξη, σύλληψη όταν έχουμε ε, δωροδοκία, όταν έχουμε διαφθορά. Ε, αυτό πάει να πει υπονόμευση της δημοκρατίας. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να ρωτηθούμε εάν το πρόβλημα είναι πραγματικό όσον αφορά την κατάχρηση των κοινωνικών πόρων. Είναι αυτό το πρόβλημα, υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις που οδηγούν σε καταφατική επάντηση. Διότι, για παράδειγμα, πριν από λίγα χρόνια η Ιταλική αστυνομία ε, μπόρεσε να μάθει ότι η μαφία ήθελε να αλλάξει τη λειτουργία της και ήθελε να καταχραστεί τους κοινούς πόρους, οπότε άλλαξε και τη στρατηγική της η Ιταλική αστυνομία. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως ας πούμε λαθρεμπόριο τσιγάρων, ε, απάτη με το ΦΠΑ, απάτη σχετικά με τις ποσοστώσεις των εκπομπών, διοξιδίου, όλα αυτά τα εγκλήματα τελούνται με διασυνοριακό έγκλημα οργανωμένο. Όπου δηλαδή αυτοί οι εγκληματίες βρουν σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2008 το Συμβούλιο είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και είχε εκδώσει σχετική απόφαση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως, το ερώτημα που αναδύεται είναι, έχουμε κάνει βήματα πρώτου, πετύχαμε τίποτα όσον αφορά το γραμμένο έγκλημα και όσον αφορά την κατάρριξη των κοινωτικών πόρων. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να συνταχθεί αυτή η μελέτη και γι' αυτό και περίμενα πώς και πώς να έρθει η μέρα για να σας μιλήσω. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο έχει πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία, χρήσιμες αναλύσεις, συστάσεις, πάρα πολύ αξιόλογες. Και δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε τους ε, συντάκτες του κειμένου. Πέραν αυτό, θα πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει κάτι που με συγκλώνησε από αυτή την έκθεση τα στοιχεία τα οποία δεν περιέχονται εδώ είναι τα πιο συγκλονιστικά που λείπουν. Αυτό φάνηκε και από την προφορική εισήγηση. Το συμπέρασμα αναφέρθηκε στο, σε σχέση με τη διαφάνεια παριθμών 13 στο τι επομένως λείπει από τη στρατηγική μας, τι δεν γίνεται. Επομένως, νομίζω ότι από πολλές πλευρές δικαιώνεται αυτό το συμπέρασμα. Άρα αυτό θέλω να δούμε. Στις σελίδες 54 και 55, πώς το λέει εδώ στα αγγλικά, λέει ότι ε, σε ποιο βαθμό γίνεται η κατάχρηση κοινωτικών πόρων σε σχέση επίσης και με το βαθμό απάτηση με ΦΠΑ για προγραμμένο έγκλημα είναι κάτι το οποίο ε, αν λάβουμε τις προφέρειες που έχουμε αυτό το ερώτημα δεν απαντάται γιατί δεν υπάρχουν αρκετέ ε, σχετικέ πληροφορίες, αρκετά στοιχεία, ε, ούτε το παρέχεται από την Όλαφη, την Europol, την Eurojust, αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο. Και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε έναν υπολογισμό ακριβή σύμφωνα με τα όσα παρατήρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι ανακοινώσει τη και επίσης ετώνησε πόσο δύσκολο είναι να έχουμε ακριβή δεδομένα για να μπορούμε να δούμε σε ποιο βαθμό να πάνε η απάτη. Δεν να υπάρχει εποπτεία, να υπάρχουν μηχανισμοί αξιολόγησης, μια που είναι αναγκαίο να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά, συνεχίζει τα σουηδικά ο εισηγητής, παρακάτω τώρα, στις σελίδες 56 και 57 πάλι στα αγγλικά αναφέρει το εξής. Σήμερα θα πρέπει να εστιαστούμε ή στα φαινόμενα της ε, επιβαρημένης περιπτώσης απάτης και εγκλημάτων και ε, στο ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία Eurojust, Europol, ε, ελεγκτικού συνεδρίου και η Όλαφ δεν προσέχει όσο χρειάζεται το οργανωμένο εγκλήμα ενώ η Europol το καταπολεμά και εστιάζει την προσοχή στην απάτη ΦΠΑ και λαθρεμπόριο τσιγάρων δεν υπάρχει άμεση ε, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Όλαφ και Europol. Ούτε υπάρχει κάποιο είδους ε, διασταύρωση στοιχείων που να γίνεται σε, σε τακτή, σε, σε μόνιμη βάση για λογαριασμού, τηλέφωνα, ε, στοιχεία ταυτότητας μεταξύ των ΜΕΝ και των ΔΕ, Όλαφ και Europol. Επομένω, δεν είναι δυνατόν να γίνουν συνδυασμοί δεν είναι εύκολο ή κάποια φορά δεν είναι αδύνατο να υπάρχει συνδυασμός και σύγκριση. Και επίσης αυτό αφορά και τον, τη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο μεταξύ αυτών των ε, φορέων και των κρατών μελών. Οπότε και δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθμό δραστηριότητας αυτών των, ε, οργανω, των οργανώσεων κλίματος και έτσι δεν μπορούμε να ενεργήσουμε τον πιο πλασματικό τρόπο. Οπότε, αυτά όλα τα οποία αναφέρει η έκθεση είναι αληθή. Και εάν είναι αληθή, είναι πάρα πολύ απογοητευτικά. Διότι δημιουργήσαμε μια εσωτερική αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα. Όμως, ταυτόχρονα, αυτό αποτελεί πεδίο δράσης των οργανωμένων εγκληματιών. Οπότε, καταλήγουμε στο ότι Όλαφ, ε, Europol, Ιούντας και λοιπά δεν συνεργάζονται, δεν συνεργάζονται αποτελεσματικά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε ούτε καν να έχουμε εικόνα της κατάστασης. Εάν λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, Και βέβαια, ελπίζω ότι κάποιος θα μου αποδείξει ότι όλα αυτά είναι αναλυθή. Εάν όμως είναι αληθή, αυτό σημαίνει ότι υπολοιπόμαστε πάρα πολύ του ευκταίου. Διότι το θέμα δεν είναι να γίνει χωροφύλακας ή κοκομπού. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, το να πιάνουμε τους εγκληματίες. Όμως, εμείς Ω πολιτική. Θα πρέπει να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα. Ποιο είναι ο υπεύθυνο, πώ μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση και έτσι θα πρέπει να διευκρινίσουμε το τι ισχύει. Και έχω όμω 10 ερωτήσει για την όλα αυτή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ελληνικό Συνέδριο. Ελπίζω ότι αυτέ οι ερωτήσει σήμερα θα βρουν απαντήσει. Πρώτα-πρώτα, ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι, γιατί να είναι τόσο δύσκολο να μπορεί κανείς να έχει μια γενικότερη έποψη του τι γίνεται του τοπίου για αυτό το θέμα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη προσβασιμότητα στα υπάρχοντα δεδομένα. Αυτά που έχουν οι επιμέρους οργανισμοί, υπηρεσίες, θεσμικά όργανα επίσης σύμφωνα με αυτήν την μελέτη δεν έχετε κάποια ενιαία συγκεκριμένη προσέγγιση πολιτική για το οργανωμένο έγκλημα. Έχετε την προσέγγιση που ισχύει για οτιδήποτε είδους έγκλημα. Άρα τι μεταβολές θεωρείτε πρέπει να γίνουν για αυτή την κατάσταση. Επίσης, άλλο, άλλη ερώτηση προς την Επιτροπή. Τι πρεσβεύεται όσον αφορά την σύσταση υπαριθμών 2, εκεί που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα, μια, ένα black list, ε, δηλαδή να είναι ένας ε, κατάλογος των προσώπων των φορέων που έχουν ε, καταχραστεί κοινωνικούς πόρους. Άλλη ερώτηση. Και στην ακρόαση και όταν πάμε από αποστολές σε διαφορετικέ χώρε, ακούμε να λένε οι δικαστέ, ότι το οργανωμένο έγκλημα καταχράται τέλος πάντων αλλοιώνει τους διαγωνισμούς για τις δημόσιες συμβάσει. Τι κάνετε γι' αυτό. Άλλη ερώτηση. Πέμπτη. Για την Όλαφ είναι αυτή η ερώτηση. Θεωρείτε ότι υπάρχει κατάχρηση κοινωνικών πόρων από το οργανωμένο στο βαθμό που αναφέρθηκε. Ή εδώ πρόκειται απλώς περί μεμονωμένων περιπτώσεων. Άλλη ερώτηση πάλι για την Όλαφ. Γιατί δεν θελήσατε ή δεν μπορέσατε να παράσχετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες στους συντάκτες αυτής της μελέτης Άλλη ερώτηση πάλι για την Όλαφ. Επί τη βάση αυτή τη και επί τη βάση των δηλώσεων τη Eurojust από ό,τι φαίνεται δεν προτίθεστε να συνεργαστείτε με τη Eurojust. Αν αυτό ισχύει, γιατί. Όγδοη ερώτηση προς την Όλαφ. Τι νομικά μέσα θα χρειαζόσασταν ούτως ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε περισσότερο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Ένα ερώτηση. το ελεγκτικό συνέδριο. Θεωρείτε ότι υπάρχει κατάχρηση πόρων από το οργανωμένο έγκλημα σε μεγάλο βαθμό. Και αν το πιστεύετε αυτό, πού το βασίζετε. Δέκατη ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο. παρακολουθείτε, εποπτεύετε το τι γίνεται όσον αφορά την, την ε, νομική, ένδικη αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις οποίες επιλαμβάνεστε. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις αν δοθούν και επίσης να ακούσουμε αντίδραση στις συστάσεις της μελέτης. Ευχαριστώ. Κυρία Ανδρέασεν, θέλει να ζητήσει τον λόγο. Θέλει κανένας άλλος το λόγο από την κυρία Ανδρέασεν. Κυρία Ανδρέασεν όμως. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τη γραμματεία και την Price Waterhouse, καθώς και τον εισηγητή για την πολύ σημαντική αυτή μελέτη. Θέλω να υποστηρίξω ένθερμα τα συμπεράσματα τα οποία κατέληξε ο κύριος Σόρενσεν και που μας παρουσίασε σήμερα. Είναι πραγματικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η μελέτη δεν μπορούσε να εξετάσει ενδελεχώς το πρόβλημα λόγω έλλειψης πληροφοριών. Ήδη αυτό είναι πολύ εύγλωτο. Μας μιλάει για τη σημασία που δίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την κατάχρηση ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω απάτης, διαφθοράς, ε, όλων των ε, αρνητικών φαινομένων γύρω από τα κοινωνικά κονδύλια. Κάτι άλλο που με ανησύχησε ακόμη περισσότερο είναι το εξή. Πριν από το συμπέρασμα για την έλλειψη πληροφοριών, είναι ορισμός του όρου κατάχρηση κονδυλίων. Αυτό με ανησυχεί. Η Pricewaterhouse ε, ορίζει την κατάχρηση ως απάτη. Αλλά πώς ορίζεται η απάτη. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον ορισμό. Άκουσα ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να ορίζει την απάντη ως κατάχρηση κονδυλίων με εγκληματική πρόθεση. Αν περιμένουμε το, ένα συνέδριο, το συνέδριο ή το δικαστήριο να αποφασίσει τι είναι δόλος, τότε θα έχουμε δυσκολίες για να διώξουμε την κατάχρηση. Ε, θα έχουμε τα χέρια μας λοιπόν δεμένα πιστάγκωνα. Δεν θα μπορέσουμε να ερευνήσουμε. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς υπάρχει εγκληματική πρόθεση. Ε, θα υπήρχαν πολύ περισσότερα δεδομένα αν υπήρχαν έρευνες ούτως ή άλλως για οποιαδήποτε παρατυπία. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μιλάει για μεγάλο αριθμό παρατυπιών κάθε χρόνο. Άρα έχουμε περιθώριο να ερευνήσουμε. Ο ορισμός της κατάχρησης των ε, πόρων είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Συμφωνώ σχεδόν με όλες τις ε, συστάσεις σας που είναι αυταπόδεικτες ε, ε, κυρίως για πολλούς από εμά αυτήν την Επιτροπή και στο, κοινο... και στο Κοινοβούλιο. Συμφωνώ απόλυτα με τη μεταρρύθμιση της Όλαφ. Συμφωνώ με την μηδενική ανοχή. Ανησυχώ για αυτή την κίνηση που γίνεται γύρω από τον ανεκτό βαθμό κινδύνου θα πρέπει να, να θεωρήσουμε την νομοθεσία για τους καταγγέλλοντες, ε, για τους αποκαλύπτοντες. Το έχουμε συζητήσει και σε μια άλλη μελέτη της Pricewaterhouse. Είναι σημαντικό. Μακάρι να είχαμε και μια, ε, ένα δεύτερο τεύχος αυτής της ε, έρευνας για όλα αυτά τα συμπεράσματα για να δούμε τι συνέχεια που σε αυτά τα συμπεράσματα. Κυρία Γκρέσλεν, καλώς ήρθατε. Είχα, συγγνώμη που άργησα. Ε, είχαμε πολλά άλλα θέματα, όπως να δούμε 500 τροπολογίες. Ευχαριστώ. Έριξα μια ματιά χθες στην έκθεση και αυτό που πρόσεξα είναι ότι η μελέτη αποκαλύπτει και πάλι τα τεράστια προβλήματα του ελέγχου των προϋπολογισμών. Δηλαδή σημαντικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Έχουμε μια βάση δεδομένων, το και Σόρεν, για να καταρτιστεί blacklist αυτό κατά χρήσης. Στον δημοσιονομικό κανονισμό του 2006 είχε αποφασιστεί μετά από αίτημα της Όλαφ να γίνει βάση δεδομένων. Αλλιώς δεν θα υπήρχε. Το Συμβούλιο προχώρησε παρά τις αντιρρήσεις οι Φιλανδοί το πέρασαν, αλλά μέχρι τώρα στην πράξη δεν λειτουργεί βάση δεδομένων. Ρωτώ την Κομισιόν λοιπόν πόσες περιπτώσεις καταγράφηκαν σε αυτή τη βάση δεδομένων. Ούτε έξι νομίζω. Άρα λοιπόν λειτουργεί το σύστημα πληροφοριών για να τροφοδοτείται και να ενημερώνει τη βάση δεδομένων, ούτω ώστε να έχει νόημα και η συγκρότησή της. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση προς εκείνους που έκαναν τη μελέτη. Η σημασία του νομικού follow-up των περιπτώσεων αυτών έχει τεράστια σημασία και είδαμε ότι πολλές φορές επειδή δεν υπάρχει νομοθεσία και δεν ορίζεται μια μορφή απάτης, δεν προκύπτει και νομικό follow-up. Εσείς τι προτάσεις θα είχατε για ένα νομικό follow-up των περιπτώσεων οργανωμένου εγκλήματος. Μετά η σύσταση υπαριθμών 8 που είναι το ε, σημαντικό. Ε, Αναφέρεστε επίσης ε, σε αυτούς που προβαίνουν αποκαλύψεις. Πώς θα επανεπεξεργαστούμε την πρόταση. Τον Ιούλιο η Κομισιόν ε, θα συζητήσει για το ε, κανονισμό του προσωπικού. Έχουμε μια ευκαιρία να παρέμβουμε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και από εσά προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε, τι θα ζητήσουμε. Άλλες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν. Καλώς τότε θα δώσω το λόγο σε τέσσερις στην Κομισιόν που θα απαντήσει σε ερωτήσεις που τους έκανε ο εισηγητής η κυρία Ανδρέασεν, η κυρία Γκρέσλε. Μετά θα δώσω τον εκπρόσωπο, ε, το λόγο στον εκπρόσωπο της Όλαφ για να απαντήσει σε ερωτήσεις που ετέθησαν σε εκείνους στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου και τέλος η κυρία Γκρέσλε ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις από τους συντάκτες της μελέτης και θα σας δώσω και σας το λόγο. Και τέλος θα έχει το λόγο ο εισηγητής, ο η Ο κύριος Φόγνας, το λέω σωστά, ο κύριος Φόγνας. Ναι, ναι, ναι, περίπου από την κυβέρνηση Διεύθυνση ε, του Υπερπολισμού έχουμε επίση εδώ πέρα και από όλε τι αρμόδιε διευθύνσει εδώ εκπροσώπου, αυτοί οι οποίοι εκταμείουν τα πιο πολλά χρήματα προ τα κράτη-μέλη και εμεί λάβαμε υπόψη αυτέ τι 10 ερωτήσει ε, που απευθύνονται στι υπηρεσίε τη Κομισιόν και ιδίω αυτέ που απευθύνονται ε, στην Όλαφ για αυτέ τι του δύο κλάδου, δηλαδή και ω ανεξάρτητη υπηρεσία που ενεργεί του Ενέργου και ω κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όμω τώρα θέλω να σταθώ στην ερώτηση παριθμών 3, η οποία περισσότερο αφορά εμάς την κυβέρνηση για τον προπολογισμό και όσον αφορά αυτή, αυτή, την πρόταση για τον blacklist, έχει δίκιο αυτό που είπε και ισχύει αυτό που είπε η κυρία ε, Γκρέσλε. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει εκτενώ όσον αφορά την, ε, τον δημοσιονομικό κανονισμό και την αναθεώρησή του και θυμάστε αυτή τη διαδρομή στηρίξαμε τις απόψεις της κυρίας Γκρέσλε και πείσαμε το Συμβούλιο που τότε είχε την απολυτική αρμοδιότητα και είχε αποδεχθεί τελικά να υπάρχει τέτοιου είδους μέτρο αποκλεισμού κλπ. Και πάρα πολλοί ήταν οι νομικοί που είχαν λάβει μέρος στην συζήτηση και είχαν πει ότι επ' αυτή τη βάση τη διαθεσμική διοργανική και εσεί με κρατημέλη δεν είναι δυνατόν έτσι να καλύψουμε όλε τι κρυθήσει υποθέσει σε σχέση με τις προσφυγές. Και επομένως, Νομίζω ότι είναι ακριβέ το που λέει η κυρία Γκρέσλε, παρά το ότι δεν ξέρω το θέμα και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και στους κόλπους της Επιτροπής έχουμε μία ούτως υπήν black list και αφορά τους άμεσα επιλέξιμους και εδώ έχουμε κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων όπου καλύπτουμε βέβαια και την απάτη. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον συνέλεγχο της Όλαφ για να απαντήσει στις ερωτήσεις που τον αφορούν. Και ό,τι δεν απαντηθεί εδώ θα το διαβάσουμε γράφος σαν απάντηση στον εισηγητή. Θέλετε και να απαντήσετε, είσαστε ο υπεύθυνο ή θέλετε τώρα να απαντήσετε ή θέλετε να, να απαντήσετε συνολικά και σε άλλες ερωτήσεις. Άρα κάποιος άλλος. Αν θέλετε όμως ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια για την πολιτική συνοχής. Περιγράφεται το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στις σελίδες 21 με 24 και θα ήθελα να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις γιατί το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει τον εποπτικό ρόλο της Κομισιόν σωστά. Κάποιες διευκρινήσεις χρειάζονται για τις εργασίες που διεξάγει η Κομισιόν τώρα. Το κείμενο ε, υπεραπλουστεύει την πραγματικότητα, πρέπει να πω, σε κάποιο βαθμό. Για την Βουλγαρία και την Ολλανδία υπάρχουν κάποιες, κάποιοι ισχυρισμοί που δεν αληθεύουν και θα ήταν χρήσιμο να είχαν ε, επικυρωθεί και διασταυρωθεί με την Κομισιόν οι σχετικές πληροφορίες. Για την Ολλανδία δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει επαρκές και σωστό follow-up στη στρατηγική ελέγχου εις ό,τι αφορά τους ελέγχους που διεξάγονται στην Ολλανδία. Η στρατηγική ελέγχου ελέγχεται κάθε χρόνο από την Κομισιόν αναθεωρείται η Κομισιόν γνωμοδοτή σχετικά με τη στρατηγική ελέγχου και τα κράτη-μέλη στέλνουν ετήσια έκθεση ελέγχου μαζί με την ε, γνωμοδότηση κάθε χρόνο που εξετάζεται από την ε, Κομισιόν. Επίσης κάνουμε συναντήσεις διμερείς για ελέγχους ε, για να δούμε τη στρατηγική ελέγχου κάθε κράτους μέλους. Η Κομισιόν επίσης κάνει δικούς της ελέγχους επιτοπίους. Για τη Βουλγαρία ε, ισχυρίζεται εδώ η μελέτη ότι η αρχή ελέγχου, η αρχή διαχείρισης και η ε, αρχή πιστοποίησης έχουν την έδρα τους στο ίδιο Υπουργείο. Αυτό δεν είναι αληθές. Στη Βουλγαρία η αρχή πιστοποίησης ε, είναι το, η Διεύθυνση Εθνικών Πόρων στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά η αρχή ελέγχου στη Βουλγαρία είναι ανεξάρτητος εκτελεστικός φορέας που λογοδοτεί στον Υπουργό Οικονομικών. Οι πέντε αρχές ελέγχου βρίσκονται σε πέντε διαφορετικούς φορείς, οπότε υπάρχει ε, σωστός διαχωρισμός των ε, αρμοδιοτήτων. Επίσης, έχουμε μια εκτενή στρατηγική ελέγχου για την περίοδο μέχρι το 2013 που στηρίζεται στην αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας. Ε, έχουμε στρατηγικές ε, πρόληψης του, της απάτης μαζί με την DGMAR, την OLAF. Επίσης κάποιες συστάσεις τώρα θα ήθελα να σχολιάσω στο τέλος της μελέτης. Εμείς ε, κάνουμε δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων και στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις επαληθεύσεις ε, διαχείρισης. Όταν πρόκειται για συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ήδη στα πλαίσια παρατυπιών και απάτης και κάθε πρόσθετες δράσεις που θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε πρέπει να γίνονται στα πλαίσια της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος και το όφελος. Είναι πολύ σημαντικές αρχές για να κρίνουμε αν θα προσθεθούν δράσεις. Οι δράσεις πρέπει να είναι αναλογικές και να λαμβάνουμε υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους. Τι θα επιτύχουμε δηλαδή με τις πρόσθετες δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις του κ. Σόντεργαρντ. Αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν τουλάχιστον κατέγραψε τις ερωτήσεις. Υπήρχαν εξάλλου ερωτήσεις που απευθυνόταν και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Θα ζητήσω λοιπόν από την Κομισιόν να απαντήσει αρκετά σύντομα στα ερωτήματα του κ. Σόντεργαρντ και αν είναι δυνατόν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος, γιατί αλλιώς ο κύριος Σόντεργαρτ θα θέσει ερωτήσεις επίσημα στο Κοινοβούλιο. Νομίζω καλό ήταν να, θα ήταν να απαντήσετε. Τέσσερις ερωτήσεις απευθύνονται προς την Όλαφ. Θα μπορούσα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Όλαφ, αν υπάρχει παρόν κάποιος, να μου απαντήσει. Ε, κύριε Πρόεδρε, είμαι υπεύθυνο για ε, το τμήμα της Όλαφ για την ε, πρόληψη της απάτης και την αξιολόγηση του κινδύνου. Λίγες παρατηρήσεις. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, η Όλαφ είναι υπεύθυνη ω ανεξάρτητο φορέα ε, έρευνας για τις έρευνες στον τομέα της καταπολέμησης απάτης και είναι και ταυτόχρονα η υπηρεσία της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μας ως ε, υπηρεσία καταπολέμησης απάτης που κάνει ε, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν διενεργούμε αυτές τις έρευνες πρέπει να σεβόμαστε τις ε, αρχές εμπιστευτικότητας κατά τις ερευνές μας. Και αν υπάρχουν πορίσματα ειδικά τα οποία προκύπτουν από τις έρευνές μας που δείχνουν εγκληματική ευθύνη, όπως παραδείγματο χάρη το οργανωμένο έγκλημα, με βάση το ποινικό δίκαιο, η Όλαφ έχει το, την υποχρέωση να υποβάλει τα αποτελέσματά στις εθνικές δικαστικές αρχές, οι οποίες ε, θα πρέπει να μπορούν είτε να διερευνήσουν, να ερευνήσουν περαιτέρω ή αν ο το θεωρήσει σκόπιμο να προωθήσει την υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια. Και αυτό εξηγεί την ε, ανάγκη να κρατήσουμε τις πληροφορίες μας εμπιστευτικές. Πρέπει να το, να το υπογραμμίσουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει απόρριτο στις έρευνές μας και να δώσουμε τη δυνατότητα να δώσουν την δέουσα συνέχεια οι δικαστικές αρχές των κρατών μεγλών. Ε, δεύτερον, ερευνούμε την απάτη, έτσι και όπως αναφέρεται στον κατάλογο του modus operandi, μερικές φορές έχουμε πλαστογραφημένα τιμολόγια ε, που δείχνουν ας πούμε κατάχρηση, υπεξαίρεση. Δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε τόσο εύκολα αυτό το, αυτά τα μόντου operandi, τον τρόπο λειτουργίας. Ούτως ή άλλως κάτι σε ερευνές μας θα πρέπει να σεβαστούμε το απόρριτο και τη δυνατότητα εμπιστευτικότητας για να έχουν περιθώρια χειρισμών οι δικαστικές αρχές. Τώρα, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε ο εκπρόσωπος ε, για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Προφανώς η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει συμπληρωματική δράση και εσείς ε, μιλήσατε για την ανακοίνωση που υιοθετήθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων μέσω του ποινικού δικαίου ε, που δείχνει σημαντικές νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Κομισιόν και ο κοινοτικός, ο ενωσιακός νομοθέτης. Θα συμπληρωθεί αυτό, αυτή η προσπάθεια από τη μεταρρύθμιση του κανονισμού 1073 Υπάρχει και ένα άλλο κείμενο που είναι σχεδόν έτοιμο να θετηθεί από την Κομισιόν και που έχει ήδη αναφερθεί από τον ε, ε, Επίτροπο που είναι υπεύθυνο ε, για την καταπολέμηση απάτης είναι η στρατηγική καταπολέμηση της Κομισιόν. Σας το έχει αναφέρει εδώ, στο Κοινοβούλιο και θα υιοθετηθεί από το Σώμα των Επιτρόπων τον Ιούνιο. Αυτή η στρατηγική Εγκολπώνται πολλές από τις σημαντικές συστάσεις που αναφέρει η μελέτη, ε, την 6, την 7 και την 8, να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για την απάτη, να υπάρχει ενίσχυση των εργαλείων για να ε, διερευνούνται οι παρατυπίες και στο οργανωμένο έγκλημα. Και μόλις η Κομισιόν ε, υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική καταπολέμηση απάτης, θα έχουμε και μια άλλη οπτική γωνία για να προωθήσουμε αυτές τις συστάσεις. Ελπίζω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Eh, Ευχαριστώ. Απαντήσατε στις παρατηρήσεις του κ. Σόντεργαρτ, αλλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη ερώτηση για την συνεργασία, η έλλειψη συνεργασίας με την Eurojust. Αυτή, σε αυτήν την ερώτηση μπορείτε να απαντήσετε. Ε, ναι, όντως, και συγγνώμη. Η συνεργασία από πλευρά Όλαφ και με την Eurojust και την Europol δεν είναι καλός. Έχουμε άμεσες επαφές και για να δούμε Πώ θα προωθήσουμε την πολιτική μα και για το πώ θα λειτουργήσουμε. Υπάρχουν τακτικέ συνεδριάσει για συγκεκριμένε περιπτώσει μεταξύ τη Eurojust και τη Όλαφ. Σε περίπτωση που υπάρχει διασυνοριακό έγκλημα και έχουμε ανοίξει διασυνοριακούς φακέλους, διασυνοριακές υποθέσει, δηλαδή, η συνεργασία είναι πολύ καλή και ελπίζω και σήμερα το απόγευμα ο Γενικός μας Διευθυντής να το επιβεβαιώσει. We zullen het εμείς θα του θέσουμε το ερώτημα, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Γκρέσλερ. Θα σα δώσω το λόγο, γιατί σα τη συγκείτε για την όλα. Ακούγοντα όλα αυτά, ε, βλέπουμε ότι δεν μάθαμε όλα όσα θέλαμε να ξέρουμε, αλλά καλό που τα συζητάμε. Αφενός έχουμε λεπτομερή στοιχεία για τις ε, περιπτώσεις απάτης και στην τελευταία έκθεση της ε, Κομισιόν είδαμε εντυπωσιακά νούμερα, στοιχεία για πρώτη φορά. Εδώ λέει ότι 0,19% των πληρωμών. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο γιατί νομίζαμε ότι θα ήταν πολύ πιο υψηλό το ποσοστό. Πάντως αυτό το 019 πώς το ερμηνεύει ο εκπρόσωπος της Όλαφ. Δεν αναφέρεται μόνο στο πρόγραμμα δράσης, αλλά είναι σαν κόκκινη κλωστή παντού, γιατί και η Κομισιόν, η Γενική Γραμματεία, έχει αρχίσει να κάνει υπολογισμούς. Και αν δούμε το PIF για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία από, χώρα σε, κάθε χώρα, ε, υπολογίζονται δηλαδή ποσοστά απάτης και υπάρχουν τρία-τέσσερα στοιχεία που παρατίθενται εκεί. Διαβάζοντάς τα είχα πάντα την εντύπωση ότι όλα αυτά ε, στοχεύουν στο να είναι χαμηλά τα νούμερα ούτως ώστε να φαίνεται μικρή η απάτη. Έχω κάποιες αμφιβολίες, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο, ποιο σωστό και ποιο δίκαιο δεν θα ήταν να λέμε, δεν ξέρουμε. Άρα τι είναι αυτό το 019. Και ξαναγυρίζω σε αυτό που είπε ο πρόσωπος της Κομισιόν. Ε, πράγματι ε, κάναμε κάποιες επίπονες μελέτες. Τώρα η Κομισιόν κάνει πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Οπότε καλό είναι να το συζητήσουμε αυτό. Η Κομισιόν λέει στην τροπολογία της ότι ακόμα και εταιρείε που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων λόγω απάτης, έχουν καταδικαστεί δηλαδή για ξέπλυμα χρήματος κλπ. Εάν έχουν ένα προϊόν ως μονοπόλιο, όλα αυτά δεν θα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, παρόλο που έχουν καταδικαστεί οι εταιρείες αυτές, ε, θα τους δώσουμε ε, ε, άφεση, για να το πω έτσι, γιατί έχουν μονοπωλιακό προϊόν. Δηλαδή, ρώτησα εγώ ποιοι είναι αυτοί και δεν μου απάντησαν. Άρα λοιπόν υποβαθμίζεται πάρα πολύ ε, η βάση δεδομένων και τα προβλήματα θεωρούνται αθώα. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε και ελπίζω, το λέω μάλιστα σκόπιμα εδώ το αναφέρω γιατί δεν θέλουμε να το ε, εξηγούμε με αφηρημένο τρόπο. Πολύ συγκεκριμένα εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα μεγάλα αυτά προβλήματα, ξέπλυμα χρήματος, ε, ε, απάτες, διαφθορά κλπ. Ναι. Όντως, δικό μας θέμα είναι, πρέπει να ασχοληθούμε. Κύριε Σόντεργαρτ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Δεν σα ακούω όμω. Να δώσουμε καταρχά το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Όχι, πρώτα στην Όλαφ, για να μιλήσει για αυτό το 0,19% που είπε η κυρία Γκρέσλερ. Όλαφ. Το 0,9% λέει ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν είναι το συνολικό ποσό στην ε, ετήσια έκθεση του Κομισιό, της Κομισιόν για το 2009-2010. Είναι όλο το ποσοστό, όλα τα ποσά απάτη σε όλους τους τομείς, ε, σε όλους τους τομείς δαπανών και βασίζεται στο ανιχνευμένο ποσοστό παρατυπιών που έχει που έχει καταχωρηθεί και για το οποίο έχει ενημερωθεί η Όλαφ από τα κράτη-μέλη. Ένας υπολογισμός που βασίζεται σε αυτή την ενημέρωση από τα κράτη-μέλη και που θα ανανεωθεί τώρα για το 2010 στην έκθεση που θα δημοσιεύσει η Κομισιόν το καλοκαίρι. Βασίζεται, επαναλαμβάνω, στο ανιχνευ... σε περιπτώσεις απάτης που αναφέρουν τα κράτη-μέλη ως ε, περιπτώσεις υπόνοιας ε, απάτης. Κάθε σωστή στατιστική έχει και ένα ε, ανεπίσημο στοιχείο. Το δηλαδή το ανεπίσημο στοιχείο, πόσο το ποσοστό μάλλον, πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι. Οι εκπρόσωποι της Όλαφ συνομιλούν μεταξύ τους. Ας τους αφήσω λίγα λεπτά να το σκεφτούν. Ίσως ο συνάδελφος, μου θα μπορούσε να μιλήσει για αυτό το, το άγνωστο, ας πούμε, ε, ποσοστό. Λέγομαι Klein Ρις. Είμαι τμήματάρχη στην Όλα και είμαι ένα από τα άτομα τα οποία συνεντευξίασε η Κούπερ για, αυτό, για αυτή την έκθεση. Ε, μετά από αυτά που ρώτησε ο κ. Σόντεργαρντ, δεν μπορώ να σας προσθέσω πολλά. Ε, δυσκολευόμαστε, το μόνο μπορώ να πω είναι ότι δυσκολευόμαστε για να καταλάβουμε το εύρος απάτης και ποιο είναι το εύρο των παρατυπιών. Υπάρχουν προβλήματα ορισμών, προφανώς. Αλλά όπως είπε η κυρία Γκρέσλερ, υπάρχουν και κάποιες ε, σκοτεινές περιοχές. Σίγουρα υπάρχει μία φαιά ζώνη, αλλά πώς ποσοτικοποιείται δεν έχουμε ιδέα. Το να πούμε ότι η απάτη είναι το 5 ή το 10% είναι υπερβολικό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί με βάση αυτά τα νούμερα προχωρούμε ούτως ή άλλως και διαμορφώνουμε πολιτικές. Και μετά, αν πούμε ένα οποιοδήποτε νούμερο τέτοιου τύπου, ας πούμε, οι πολιτικές θα ήταν δυσανάλογες, θα ήταν α, λάθος, ας πούμε. Φυσικά, οι ερευνητές θα ήθελαν να γνωρίζουν το έύρο του φαινομένου και δεν το γνωρίζουν, αυτό τους δημιουργεί απογοήτευση, αλλά και εμείς αντιμετωπίζουμε την ίδια ακριβώ απογοήτευση με τους ερευνητές. Ευχαριστώ. Το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί υπήρχαν δύο ερωτήματα που αφορούσαν συγκεκριμένα το ελεγκτικό συνέδριο. Κάτι την απόψή σα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα, τι, απάτη, τι απάτες κάνει, τι... Μπορείτε να μας δώσετε κάποια νούμερα, μπορεί να απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήρθα για άλλη δουλειά, αλλά παρεμπιπτόντως μου φάνηκε ενδιαφέρον και θα σας τα πω. Οπότε, σας τονίζω ότι η έλεγχη μας λαμβάνει υπόψη το στοιχείο της ε, απάτη σαν ε, ρίσκο, ακριβώς όπως το είπε ο πρόεδρος στις 15 Απριλίου στην επιστολή του. Αυτό Αυτοδικαίω εξετάζεται. Επίση το θέμα είναι κατά πόσο θεωρούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένας μεγάλος βαθμός εκτεταμένε πάντας σε διάφορου τομεί όσον αφορά του τους ε, πόρου, α ας πούμε την περίπτωση την υπόθεση καρουσέλ και εκεί πέρα ξεκάθαρα ορίζεται ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Επομένω έγινε αυτό. Επίση τώρα να επανέλθω σε μία από τι ε, συστάσει τη έκθεση εκεί όπου ακριβώς όπω είναι διατυπωμένο, νομίζω ότι θα προκαλέσει προβληματισμό, διότι εδώ μιλά για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Όλαφ και Αλληλεγκτικού Συνεδρίου. Εάν ο ελεγκτή ανοιχνεύσει απάτη, τότε κάνει πάσα την υπόθεση στους αρμόδιους για τις έρευνες και λέμε ότι όσο περισσότερο το ψάξουμε για την αστυνομική, ενδεχομένως αυτό να είναι στοιχείο εμπλοκής για την ποινική δίωξη. Άρα παραπέμπουμε την περίπτωση στην Όλαφ. Επομένως, έτσι το βλέπουμε. Δεν προσδοκούμε τίποτα πληροφορίες από την Όλαφ όσον αφορά φερόμενες υποθέσεις απάτες που εκείνοι ερευνούν, διότι θεωρούμε ότι από τη μία έχουμε την υποχρέωση διαφάνειας και από την άλλη την υποχρέωση απορρίτου. Είναι απαραίτητη για να έχουμε μία δίκαιη δίκη, να έχουμε την υποχρέωση της, του απορρίτου. Τώρα, αν παρακολουθούμε την εξέλιξη των υποθέσεων, ναι, έχουμε σε τακτά διαστήματα συναντήσεις με την Όλαφ, και όταν παραπέμπουμε υπόθεση σε αυτούς, δεν κλείνει το θέμα για μας, γιατί σχεδόν πάντα η Όλαφ επανέρχεται, μιλά με τους ε, ελεγκτές, ε, μελετούν τους φακέλους, οπότε έχουμε συνεχή επαφή με την Δεν ξέρω αν έχουμε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το πόσες υποθέσεις κατέληξαν σε, σε έγκυρες ποινικές διώξεις, αλλά θα το δούμε. Ευχαριστώ. Για ναι. μου, όταν ε, ασκείται κάποιον τον έλεγχο και υποψιάζεται ότι υπάρχει στοιχείο απάντηση και το παραπέμπεται αυτό στην όλα αυτό που μας είπατε. Για πετε μας, αυτό πόσο συχνά συμβαίνει. Συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Έτσι μπορεί να μας πείτε ένα ποσοστό. Είναι κάτι που σημαίνει κατεξαίρεση. Μπορείτε να μας πείτε. Ο πρόεδρος Εμιστολή είπε ότι έχουμε περίπου τρεις υποθέσεις ετησίως. Καμιά φορά τα κρατημέλη ειδοποιούν για κάποια υπόθεση την Όλαφ. Δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Αλλά όταν εμείς ασκούμε έλεγχο έχουμε μια που ελέγχουμε χιλιάδες συναλλαγών έχουμε τρεις υποθέσεις ετησίως. Ευχαριστώ. Δηλαδή, είναι νομικά υποχρεωτικό να ενημερώσετε την Όλαφ για, τέτοια, για τέτοιες περιπτώσεις ή είναι δυνητική αυτή η δυνατότητα. Πολύ καλή ερώτηση. Είναι μέρος του κανονισμού μας αυτό. Όλοι οι ελεγκτές έχουν τις ε, οδηγίες τους. Ίσως η Όλαφ μπορεί να μας ε, ε, πει εάν πρόκειται για νομική υποχρέωση, αλλά εμεί το κάνουμε. Νομίζω ότι η νομική βάση είναι ο κανονισμός 1073 που λέει ότι στο άρθρο 7 ότι όλα τα θεσμικά όργανα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να υποβάλουν εκθέσεις για σοβαρές ε, υποψίες ε, παρατυπιών και να τις αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ. Είχε γίνει και μια ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε για τους συντάκτες της έκθεσης δεν τη θυμάμαι εγώ, αλλά θα τη θυμάστε εσείς, είμαι βέβαιος. Για το κανονισμό του προσωπικού και τις συστάσεις μας. Ε, θέλω να αναφερθώ σε μια άλλη μελέτη που κάναμε και παρουσιάσαμε εδώ ως PricewaterhouseCooper με κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τους ε, προβαίνοντες σε αποκαλύψεις. Ε, υπάρχουν, είπαμε, κάποια άρθρα που αποθαρρύνουν ε, τις αποκαλύψεις και είπαμε ότι ίσως τα άρθρα αυτά είναι περιορισμένα και προτείναμε γι' αυτό να αναδιατυπωθούν τα σχετικά άρθρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην άλλη έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει εδώ στο Κοινοβούλιο. Επίσης για τον ορισμό, τον νομικό ορισμό της απάτης, είχαμε βέβαια δυσκολίες να καταλήξουμε σε έναν ενιαίο ορισμό της απάτης, όμως υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που καταγράφουμε στην έκθεσή μας επίσης, που μπορούν να θεωρηθούν ως συμπεριφορές ε, που οδηγούν σε απάτη, δόλιες συμπεριφορές. Αλλά είναι δύσκολο να έχουμε έναν ορισμό μόνο. Ίσως εδώ μπορούν να βοηθήσουν οι οργανώσεις πολέμηση της απάτης, όλα κλπ. Δεν κάναμε δηλαδή μια κανονική νομική μελέτη σχετικά με τους ορισμούς και πώς μπορούν να τροποποιηθούν ε, εμείς ε, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το στάδιο το κάναμε και το καταγράψαμε. Ευχαριστώ. Ας δώσουμε το λόγο τώρα στον ε, κύριο Ζόντεργκάρτ για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Κατανοούμε βεβαίως ότι δεν είναι όλοι εις θέση να απαντήσουν έτσι άμεσα σε όλες μου τις ερωτήσεις. Θα είμαι πολύ ευτυχής αν ε, αργότερα πάρω τις απαντήσεις σας. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτό το σημείο για τη σαφή θέση τους σχετικά με την κατάχρηση των ε, ενωσιακών πόρων, πώς ε, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Η Όλαφ όμως δεν ήταν εξίσου σαφής ε, επ' αυτού. Η Όλαφ πιστεύει ότι οι προσπάθειες κατάχρησης των πόρων της Ένωσης είναι ένα πρόβλημα κοινό ή μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση για αρκετούς λόγους. Καταρχήν, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε, μίλησε για την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους, γιατί δεν πρέπει να δαπανούμε υπερβολικούς πόρους για κάτι που δεν συνιστά ίσως τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε κάποια ανεπίσημα ε, στοιχεία αλλά πρέπει να έχουμε μια εκτίμηση σχετικά με την τάξη μεγέθους του προβλήματος, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι ότου συντελεστεί ε, η απάτη. Πρέπει να ξέρουμε για ποια ποσά μιλάμε, για να μπορούμε να ξέρουμε τι ποσά θα δαπανίσουμε για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μας πείτε, είναι μεγάλο πρόβλημα ή κάποιες ε, διάσπαρτες μεμονωμένες περιπτώσεις. Επίσης, το διασυνοριακό ε, οργανωμένο έγκλημα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο προκαλεί μεγάλη ζημιά. Δεν πρόκειται μόνο για μια μικρή απάτη, γιατί το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα μπορεί να επηρεάσει και τη λήψη των αποφάσεων, πολιτικών και διοικητικών. Και εκεί είναι ο μεγάλος ο κίνδυνος Μιλάμε για χρήματα βέβαια. Τα χρήματα ε, μπορεί να είναι πολλά και να δημιουργούν πρόβλημα, αλλά το ουσιαστικό πρόβλημα είναι όταν ισχυροποιηθούν τόσο πολύ οι εγκληματικέ οργανώσει ώστε να επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων πολιτικών, διοικητικών. Είναι ένας κίνδυνος αυτό σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άγνωστες παράμετροι, αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουν για να έχουμε κάποια σαφή εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος, για να ξέρουμε ε, κατά συνέπεια πόσους πόρους θα χρειαστεί να δαπανίσουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να πω επίσης ότι εξακολουθώ να αισθάνομαι κάποια σύγχυση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να έχουμε μια εποπτεία αυτού του προβλήματος. Σέβομαι το θέμα της εμπιστευτικότητας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Καταλαβαίνω τη θέση της Όλαφ πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν ζητάμε να αποκαλυφθούν ονόματα όμως Οι συγκεκριμένες μέθοδοι ε, διάπραξης της απάτης για να φωτιστούν κι άλλοι. Ε, αυτά πράγματι πρέπει να είναι στοιχεία που θα τα προστατέψουμε. Εδώ στο Κοινοβούλιο όμως έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πόσα περιστατικά έχουν εντοπιστεί. Ε, σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να δοθεί συνέχεια γιατί αν δεν έχουμε ποπτία της κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να ε, λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις για τη λύση του προβλήματος. Πάντως, σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας και θα περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις της εκρεμής ακόμα ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια θα κλείσουμε με το σημείο αυτό φτάνοντας έτσι και στο τέλος της πρωινής μας συνεδρίας. Τώρα κάποια πρακτικά θέματα. Στις 5.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές, οπότε φροντίστε να αρχίσουμε με ακρίβεια. Το πρώτο τέταρτο θα μιλήσουμε για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με υποβολή εκθέσεων και στις 6 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι είναι μεγάλο το διάλειμμα όχι για την κυρία Γκρέσλε που θα εξετάσει 482 τροπολογίες αλλά θα, έχουμε, θα επανέλθει στις 3 με 4 για να έχουμε την κοινή συνεδρίαση ε, Κοκομπιού και ε, Επιτροπής Προϋπολογισμού ε, και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.